και 9 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται ε, 124 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται 126 υπέρ 27 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές έγκρινεται 131 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται 128 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται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 αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές Α, δεν κατάλαβα. Ε, ηλεκτρονικός έλεγχος. Για την 17β, τροπολογία 4. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 24 ψήφους κατά και 4 αποχές. Τώρα έχουμε την γνωμοδότηση της Περιφερειακής Επιτροπής. Και περνάμε στην τροπολογία Reggie 4, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Reggie 6, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Υπάρχουν ακόμα τρεις που αν συμφωνείτε, η Reggie 6, 7, 8, 9, να τις ψηφίσουμε από κοινού. Ωραία λοιπόν, τις τρεις που είπα, 7, 8, 9, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Πάμε τώρα στην ε, Επιτροπή Εμπορίου, ίντα 1, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τώρα, στην Ήτρε 3 και 4, αν συμφωνείτε, τις ψηφίζουμε από κοινού, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Μπορούμε να προτείνουμε επίσης για εδώ ψηφοφορία unblock για όλες τις τροπολογίες της ΣΥΤΡΕ, δηλαδή 6, 8, 10, 11, 12, 15. Όχι, δεν συμφωνείτε. Ωραία, μία προς μία. Ήτρα 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Εγκρίνεται. Ήτρα 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ήτρε 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ήτρε 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ήτρε 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ήτρε 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ήτρε 17 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Ήτρε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21 Ήτρε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Πάμε στην 24 ή 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά άρχεται η 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Chiusa la votazione. Τέλος της ψηφοφορίας. 44 υπέρ 0 κατά. 6 αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Γκουρεάνο. Εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία procediamo ora alla votazione del rapporto dell'onorevole eh, Galler su eh, una eh, politica sostenibile per la... Έχουμε την έκθεση του κυρίου Γκάλερ για την βιώσιμη πολιτική της ΕΕ για το Βόρειο Πόλο. Περνάμε στην τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 41, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ, συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε λοιπόν στην τροπολογία 48. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 50. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 51. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 52. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 53. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε στην τροπολογία 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Αποσύρεστηκε το 66 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 69 ε, ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 71 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται συμβιβαστική 5 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 77 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 78 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 79 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 80 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 81 και 84 είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται προφορική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε στην 87 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και περνάμε στην τροπολογία 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Πάμε στην 99. 99 που είναι συμβατή με την 8. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 102. Α, θέλετε να ελέγξουμε την 99. Ελεκτρονικά, κόσα έλεγχος της 99, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. 25-25. Απορρίπτεται. 102. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αλλά δεν είμαι βέβαιος λοιπόν ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά το 112 Τέλος της ψηφοφορίας. 32 ναι, 21 όχι. Εγκρίνεται. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 116 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 117 υπέρ κατά ε, δεν καταλαβαίνω ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την 117 σας παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια γιατί μετά χάνουμε χρόνο με την ηλεκτρονική ψηφοφορία 53 50... 40 κατά, 13 υπέρ, απορρίπτεται. Δεν σηκώσατε τα χέρια. Λοιπόν, 118 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 19, 119 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 121 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 122 υπέρ. Κατά Πάλι δεν βλέπω. Νομίζω πως απορρίπτω, αλλά δεν είμαι σίγουρος. 122 λοιπόν, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε. Chiusa la votazione. Τέλος ψηφοφορίας. Ε, τι θέλετε τώρα δηλαδή. Με κορυδεύετε. 43 <laughs> κατά, 8 υπέρ. Μα είναι τεράστια πλειοψηφία. Θέλετε να με κουράσετε. Αν με κάνει θα δουλέψω περισσότερο από σήμερα. Bon, ας πάμε στην 123 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 124 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 125 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 126 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 127 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται προφορική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 128 με προφορική τροπολογία του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 131 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, ε, συμβαστική 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στη συμβιβαστική 11, ποιοι είναι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβιβαστική 13, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 141, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 142 υπέρ κατά εγώ νομίζω πως απορρίπτεται εντάξει ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικός έλεγχος ε, ναι, αυτές οι αβεβαιότητες τι να κάνουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με δύο ψήφους παραπάνω. Εντάξει, εδώ ήταν δύσκολο. Όντως εγκρίνεται. 142 ήταν αυτή. Πάμε τώρα να ψηφίσουμε την 143. Υπέρ. Κατά. πουχές απορρίπτεται. 144 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 146 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 147 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 149 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 148 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 150 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 151 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 154 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 153 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 150, 161 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 162 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 163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 αποχές απορρίπτεται 31 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2-3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 4 κάθετος 6. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θα σας πρότεινα τις 8, 9 και 10 να τις ψηφίσουμε από κοινού αν δεν έχετε αντίρρηση. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 11. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 13. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελικό ψήφισμα ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας Ομοφωνία ούτε μία ψήφος κατά, 46 υπέρ, 7 αποχές, συγχαρητήρια. Κύριε Σιγητά, εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία. Μπράβο κύριε Γκάλερ. Μια στιγμή να συμβουλευτώ εδώ τη γραμματεία. Bene, Καλώς. Περνάμε στην, έκθεση για τις διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Λιβύης. Η συγκίτρια κυρία Γκόμες, 25 έχει αποσύρθει, οπότε ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία 1 της συγκίτριας. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 26, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 31. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 32 υπέρ ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 31 άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέλος, 25 είπα ναι και 26 όχι, άρα απορρίπτεται. Τροπολογία 32, ποιος είναι υπέρ. Κάποιος ζήτησε το λόγο. Παρακαλώ, μετρήστε και τη δική μου ψήφο υπέρ, γιατί έκανα λάθος το κουμπί. Μία επιπλέον ψήφος δηλαδή υπέρ. Αλλά δεν αλλάζει τίποτα ούτε με τη δική σας ψήφο, γιατί από τη στιγμή που έχει σοπαλία απορρίπτεται. Ένα καφέ παρακαλώ στον συνάδελφο για να ξυπνήσει. Την 31 την ψηφίσαμε. 32. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 35 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 36 υπέρ, 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές Α, δεν είναι σίγουρο για την 39 ηλεκτρονική ψηφοφορία αρχιτή ψηφοφορία Τέλος. Τριάντα υπέρ, 21 κατά, μία εποχή, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 46 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 47 λέει πάλι ο πρόεδρος. Υπέρ. Κατά. δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε την 47 ηλεκτρονικά. Άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Με μία ψήφο διαφορά όντως ήταν οριακή ψηφοφορία. Απορρίπτεται 48 υπέρ, κατά, αποχές. Ούτε και εδώ είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονικός έλεγχος λοιπόν για την τροπολογία 48. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Και πάλι οριακά 26 με 27 για μία ψήφο διαφορά απορρίπτεται. Άρα περνάμε στη 49. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 50. Θέλετε και πάλι επαλήθευση για τη 49. Εντάξει, αφού το ζητάτε θα το κάνουμε. Χάνουμε χρόνο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 49. 49 τέλος ψηφοφορίας 24 υπέρ 28 κατά απορρίπτεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές μάλλον εγκρίνεται αλλά δεν είναι βέβαια 100%. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 51. Παρακαλώ, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος η ψηφοφορία. 27 υπέρ, 25 κατά εγκρίνεται. Αλλά πραγματικά στην κόψη του ξεραφείου. 52 ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, Ούτε και εδώ είναι σαφέ το αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για την 52. Ψηφίσατε όλοι, τέλος. Εγκρίνεται και πάλι με δύο ψήφους διαφορά, 26 προς 24. Ψηφίζουμε την 53, ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 55, ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές Απορρίπτεται. 58. Γιατί εγκρίναμε την 55, την απορρίψαμε, άρα να ψηφίσουμε την 56, εντάξει. 56, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 57, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 58 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 60 υπέρ κατά αποχές μάλλον απορρίπτεται η 61 έχει αποσυρθεί συμβαστική τροπολογία 4 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται περνάμε στην τροπολογία 10 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Μάλλον απορρίπτεται. Αλλά δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά. Ας ψηφίσουμε το 11. Τροπολογία 11 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 11. Τέλος ψηφοφορίας. 23 ψηφί υπέρ, 29 κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα γι' αυτό θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για τη 17 άρχεται η ψηφοφορία τροπολογία 17 τέλος ψηφοφορίας με μία ψήφο διαφορά εγκρίνεται πώς να καταλάβω 26 υπέρ 25 κατά Οριακά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Μάλλον απορρίπτεται. Αλλά στο ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Ξέμεινε κανένα όχι. Τέλος ψηφοφορίας. 25 υπέρ, 27 Κατά. Απορρίπτεται. 19. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Μάλλον η ίδια κατάσταση. Αλλά στο απαληθεύσουμε και ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για το 19. Τέλος της ψηφοφορίας. 24 προς 29 απορρίπτεται. Ποιος είναι υπέρ του 20. Κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι σαφέστερο το αποτέλεσμα. 21 καθέτος 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 24 είναι συμβατή. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τρία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τέσσερα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πέντε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελικό ψήφισμα ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας κάποιος χρειάζεται καφέ επιγόντως Συγχαρητήρια, Παμψηφί! 52. Θρίαμβος, θρίαμβος κυρία Γκόμες. 52. Λοιπόν, μια τεχνική σφίσης παύση, διάλειμμα για 5 λεπτά και μετά θα προχωρήσουμε στην υπόλοιπη ψηφοφορία. Κοιτάξτε, βγάλτε τις κάρτες τώρα από τη σχισμή γιατί μετά θα τις ψάχνετε. Ε, Συνάδελφοι, παρακαλώ. Please, colleagues, we have to start. To start, uh, the time is uh, limited. Πρέπει να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρέπει να συζητήσουμε την πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την έκθεση πρόοδου της Τουρκίας. Η συγκίτριά μας, κυρία Μανερά, να σβιαστεί να καθίσει για να ξεκινήσει την παρέμβασή της. Καρά, της αφήσω δύο λεφτά για να κάτσει. Και έχουμε κάποιες υποδείξεις να σας κάνουμε πριν να ξεκινήσει η συζήτηση. Να σας θυμίσω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών έχει οριστεί για τις 10 Ιανουαρίου 2011. Και έπειτα θα εξετάσουμε εκ νέου το σχέδιο ψηφίσματος για την συζήτηση των τροπολογιών την 1η Φεβρουαρίου. Η τρίτη λοιπόν εξέταση και ψηφοφορία στην Επιτροπή προβλέπεται για τις 10 Φεβρουαρίου. Λοιπόν, αφού σας τα είπα όλα αυτά, να δώσω το λόγο για 5 λεφτά στην εισηγήτρια Όμεν Ρόιτεν. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ και μερικές ημέρες έχετε πάρει την ε, νέα έκθεση την οποία και κατάρτισα βάσει της εκτέσεις προοδού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά, Πρόεδρε, έκανα και πάρα πολλές συζητήσεις, όχι μόνο στις Βρυξέλλες, αλλά και στην Τουρκία. παρακολούθησα και πολύ τον τύπο στην Τουρκία και χαίρομαι και θεωρώ τιμή μου που σας υποβάλλω σήμερα το σχέδιο έκθεσης αυτής. Ξέρετε ότι πάντα προσπαθώ να μην τονίζω μόνο τις αρνητικές εξελίξεις, αλλά και τα θετικά στοιχεία. Αυτό το κάνω κατονομάζοντας και κάποιες προτεραιότητες. Στην προηγούμενη, στις προηγούμενες εκθέσεις μου πάντα ανέφερα ότι το πιο σημαντικό θεωρώ σε ό,τι αφορά τη συνεργασία και την πρόοδο του φακέλου της Τουρκίας είναι τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Και γιατί? Γιατί πρόκειται για τον πυρήνα, την καρδιά της συνύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όποιο θέλει να προσταθεί σε αυτήν πρέπει να πληρεί τα κτίρια αυτά. Πρόκειται για τη δημοκρατία, τα ε, δικαιώματα των πολιτών, το κράτος δικαίου με ανεξάρτητη και μερόληπτη ε, δικαιοσύνη. Πρόεδρε, αυτά μας ενώνουν στην Ευρώπη και αυτά θα πρέπει να πληρούν οι υποψήφιες χώρες. Και αυτό εξακολουθεί να αποτελεί τη δική μου προτεραιότητα. Και θεωρώ ότι για μια χώρα όπως την Τουρκία είναι πολύ σημαντικότερο να συνεργάζεται και να εργάζεται καλά για τα πολιτικά κριτήρια από το να εργάζεται για κεφάλαια τα οποία μπορεί και να μην υπάρχουν. Και η Κύπρος, αν ε, επιληθεί το Κυπριακό, θα ανοίξουν και πιο πολλά κεφάλαια. Πρόεδρε, είναι πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των πολιτικών κριτηρίων, θα πρέπει να υπάρξουν λοιπόν μεταρρυθμίσει στη χώρα. Και οι μεταρρυθμίσεις στη χώρα αποτελούν το πρώτο θέμα που επιλέγω να τονίσω. Μιλάμε για την ε, πόλωση η οποία εξακολουθεί να υφίσταται σε κάποιους τομείς. Τεράστια πόλωση μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, των ε, διοικητικών υπηρεσιών αλλά και στο εσωτερικό της κοινωνίας και αυτό εμποδίζει τις μεταρρυθμίσεις για τον περαιτέρω εκδημοκρατισμό και εκμοντερνισμό της τουρκικής κοινωνίας θα πρέπει να υπάρξει προθυμία για την εξέβρεση συνένεσης και συμβιβασμών και θεωρώ ότι η τουρκικό κοινοβούλιο θα πρέπει να παίξει σημαντικότερο ρόλο. Αλλά θεωρώ, Πρόεδρε, και αυτό είναι καινούργιο και το αναφέρω τέσσερις φορές στην έκθεση, θα πρέπει να υπάρχουν πιο πολλά θέματα ε, ελέγχων και ισορροπιών. Θεωρώ ότι τα κόμματα θα πρέπει να συνομιλούν μεταξύ τους. Δεν είναι δυνατόν ένας να κερδίζει τα πάντα. Θα πρέπει σε διαπραγματεύσεις, θα πρέπει να υπάρχουν δυνατότητες ε, και για την αντιπολίτευση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το checks και balances ε, στην κοινωνία και στο κοινοβούλιο ιδιαίτερα θα πρέπει να λεφθούν περισσότερο υπόψη. Δεύτερο σημείο, σημείο συστηματικές μεταρρυθμίσεις. Είπα και το προηγούμενο έτος ήμουν πολύ ενθουσιώδης για το δημοκρατικό άνοιγμα Μία προσέγγιση η οποία ε, θέλαμε να συμβεί προς όλες τις θρησκευτικέ κοινότητες, στους Αλεβίτες και προς τους ε, Κούρδους. Τότε το είχα χαιρετήσει. Και τι βλέπω τώρα, Πρόεδρε, ότι με τις λέξεις, θεωρητικά, πολλά συμβαίνουν. Και είμαστε ευγνώμονες για πολλές στατικές χειρονομίες που έχουν λάβει η χώρα. Αλλά δεν υπάρχει συστηματική ε, παρακολούθηση των πρωτοβουλειών αυτών. Άρα ζητώ στην έκθεση να υπάρξει συστηματικότητα σε ό,τι αφορά το δημοκρατικό άνοιγμα, τη συμμετοχή όλου του πληθυσμού στην τουρκική κοινωνία. Πρόεδρε, επιπλέον, εξακολουθούν να υφίστανται προβλήματα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας και αυτό σε πολύ σημαντικούς τομείς πολύ καλή νομοθεσία σε πολλού τομεί, αλλά όχι η εφαρμογή τη νομοθεσία. Και αυτό πρέπει να συμβεί. Τώρα, για τη συνταγματική αναθεώρηση, Πολλέ φορέ το έχουμε συζητήσει, έχουμε διαπιστώσει ότι τα κεφάλαια τα οποία πήγαν σε δημοψήφισμα ήταν ένα καλό βήμα προς ε, τη σωστή κατεύθυνση, αλλά σε τελική ανάλυση θα πρέπει να υπάρξει μια συνολική συνταγματική αναθεώρηση. Και στην τελευταία μου επίσκεψη μίλησα με την ε, αντιπολίτευση και κατάλαβα ότι και εκεί υπάρχει η αντίληψη ότι θα πρέπει να υπάρξει συνταγματική αναθεώρηση για τη συστηματική αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ελπίζω μετά τις εκλογές να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό. Τώρα, Πρόεδρε, Υπάρχουν και κάποια θετικά στοιχεία τα οποία θα ήθελα να αναφέρω ιδιαίτερα. Θεωρώ ότι υπάρχει πιο μεγάλος έλεγχος ε, στο στρατό. Άλλα καινούργια στοιχεία για την ελευθερία του τύπου. Ανησυχώ για την αυξανόμενη πίεση στον ε, τύπο, στην ελευθερία του τύπου και σε ό,τι αφορά τη λογοκρισία. Είχαμε το άρθρο 301 το οποίο και προσαρμόστηκε και αυτό φαίνεται ότι λειτουργεί, Πρόεδρε. Είχαμε κάποια ερωτηματικά, αλλά εν πάση περιπτώσει λειτουργεί. Τώρα όμως τι βλέπουμε, ότι με αποποίηση των αρχών και από το δικαστικό κλάδο έχουμε όλο πιο, πιο πολύ αυτολογοκρισία, πολύ επικίνδυνο αυτό και να συμφωνήσω με τον πρόεδρο Γκουλ που είπε ότι στη δημοκρατία είναι σημαντικό, απαραίτητο να υπάρχει πλουραλισμός των μέσων και ελευθερία του τύπου. Πρόεδρε, ε, δίνω ιδιαίτερη σημασία στη θέση των γυναικών. Επικεντρώθηκα στο θέμα αυτό. Γίνεται πάρα πολλά για την εκπαίδευση των νεαρών κοριτσιών και γυναικών, αλλά διαπιστώνουμε ότι έχουμε 200.000 κορίτσια που δεν πηγαίνουν στο δημοτικό. Θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Αναφέρω επίσης θέματα ε, εγκλημάτων τιμής. Ε, καλή είναι η νομοθεσία, όχι όμως η εφαρμογή. Επισκέφθηκα και κάποια καταφύγια, κάποια κέντρα για τέτοιες γυναίκες, τα οποία είναι πολύ περιορισμένα αριθμό. Δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία και για παράδειγμα, στα καταφύγια μπορεί να μείνει κάποια κοπέλα μόνο τρει μήνε και μετά την αναγκάζουν χωρί μέσα να επιστρέψει στα άτομα τα οποία ε, είχαν εγκαταλείψει. Εδώ λοιπόν κάτι πρέπει να γίνει. Τέλος, Πρόεδρε, γιατί με κοιτάτε επίμονα. Θέματα βιώσιμη ε, κοινωνίας. Στην το τελευταίο δημοψήφισμα δόθηκαν ε, επιπλέον δικαιώματα και στα συνδικάτα. Ζητώ λοιπόν επανειλημμένα από την Τουρκία, από την τουρκική κοινωνία να ε, δεσμευτεί υπέρ του πολιτικού διαλόγου. Γιατί θα πρέπει οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι, οι μικρές, οι μεγάλες επιχειρήσεις ε, να μπουν σε ένα πολιτικό διάλογο, σε ένα κοινωνικό διάλογο. Πρόεδρε, ανησυχώ σε ό,τι αφορά την νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντο και διάφορε μη κυβερνητικέ οργανώσει έχουν επιστήσει την προσοχή μα σε αυτό, το διαπίστωσα και εγώ. Ο συνήθως το συμπληρωματικό πρωτόκολλο και το κυπριακό. Δεν έχω αλλάξει το κείμενό μου στο θέμα αυτό. Είναι ακόμα πιο κατεπήγον το θέμα γιατί αφορά και κάποια ε, κεφάλαια σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική. Η Τουρκία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην περιοχή. Καλές εξελίξεις, αλλά ζητώ πολλά παραπάνω, πολύ περισσότερο συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ευθύνε εδώ. Αυτά, Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι σημαντικό όπως κάναμε και τα άλλα χρόνια, να προσπαθήσουμε να περιοριστούμε σε ό,τι αφορά την κατάθεση τροπολογιών, γιατί αυτές, ξέρετε, αποδυναμώνουν το μήνυμα. Θα ήθελα λοιπόν να μην έχουμε πάρα πολλές τροπολογίες και καλό τους συναδέλφους να συνεργαστούν. Θα διαπραγματευτώ και με τους ε, σκιώδεις για να είναι ε, ευρία η αποδοχή της έκθεσης αυτής από το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ευχαριστώ κυρία Ξεκινάμε με τους όδους εισηγητές. Δύο λεπτά, ο κύριος Ομπιόλς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Διάβασα με ιδιαίτερη προσοχή την έκθεση της κυρίας Όμεν Ρόιτεν και πιστεύω ότι είναι πολύ αξιόλογο το έγγραφο. Καταβάλει προσπάθειες να συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως προς την πρόοδο που έχει επιτελέσει η Τουρκία στην ε, ενταξιακή της διαδικασία. Και φυσικά θα εξετάσουμε την έκθεση με ιδιαίτερη προσοχή. Θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε τη σύστασή της και να μην το παραξηλώσουμε στις τροπολογίες. Πάντως πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε έμφαση σε κάποια σημεία. Τα έθιξε κάπως η συγγήτρια. Για παράδειγμα, την ανάγκη η μεταρρυθμιστική διαδικασία στην Τουρκία να συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση και να υποστηριχθεί από το πολιτικό φάσμα, από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, αλλά και από σύσσωμη την τουρκική κοινωνία. Οι μεταρρυθμίσεις προχώρησαν κατά τη διάρκεια του 2010. Είχαμε τη συνταγματική αναθεώρηση καταρχήν. Αλλά το να κρίνουμε θετικά την συνταγματική αναθεώρηση, ναι μεν καλό είναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι δεν υπήρχε συμφωνία κυβέρνηση και αντιπολίτευση και δημιουργήθηκε αδυναμία ως προς την διεκπαιρέωση των εξυγχρονιστικών και προοδευτικών μεταρρυθμίσεων της χώρας. Θα ήθελα τέλος να ζητήσω από την Προεδρία αν γίνεται να παρατείνουμε κατά μία εβδομάδα τη διορία για τις τροπολογίες. Αν δεν κάνω λάθος, λίγη η προθεσμία στις 10 Ιανουαρίου, που είναι η πρώτη μέρα ουσιαστικά ε, δραστηριοτήτων, επανάληψη των εργασιών μετά τις χριστουγεννιάτικες διακοπές, θα προτιμούσα μία εβδομάδα επιπλέον. Καλώς, θα εξετάσουμε την πρότασή σας, θα δούμε αν ε, είναι εφικτή. Ο κύριος Λάμσδορφ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ρία Ράιτον για τη συνηθισμένη ε, καλή της εργασία σε ό,τι αφορά το σχέδιο έκθεσης. Νομίζω ότι στο αιτιολογία Α αποτυπώνεται η συνένεση που επικρατεί στο Κοινοβούλιο ε, σε ό,τι αφορά το ανοιχτό τέλος των διαπραγματεύσεων μιας δύσκολης διαδικασία για την ένταξη. του κείμενο σε ορισμένες ε, περιπτώσεις είναι πολύ επικριτικό και νομίζω ότι αυτό ορθώς και είναι έτσι. Από φιλελεύθερης πλευράς ε, πρέπει να πω ότι ευχαριστώ ιδιαίτερα την ε, συνάδελφο που θίγει το θέμα της ελευθερίας του τύπου σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των κριτηρίων της Κοπενχάγης. Είναι βασικό το θέμα αυτό για μας και το θέμα της αυτολογοκρισίας που αναφέρεται. Μας ανησυχεί ιδιαίτερα ότι υπάρχουν για παράδειγμα μποϊκοταρίσματα του Πρωθυπουργού εναντί κάποιων μέσων ενημέρωσης, εναντί κάποιων εκδοτών, κάποιων εφημερίδων που ασκούν ε, κριτική στην ε, κυβέρνηση. Και αυτό ε, καταδεικνύεται ότι δεν είναι θετικέ οι εξέλιξει στο σημείο αυτό στην Τουρκία. Σε ένα σημείο πρέπει να πω ότι είμαι απαγοητευμένο, ιδιαίτερα απογοητευμένο εδώ και χρόνια έχουμε συζητήσει ε, με του συναδέλφου από την Τουρκία Εθνοσυνέλευση και πάντα αναφέρεται το θέμα του 10% ε, του ορί του 10% για την είσοδο στο κοινεβόλαιο. Στο Κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη χώρα στον ΩΣΑ που να έχει τόσο υψηλό ποσοστό χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση και θεωρώ ότι σωστή είναι η έκκληση προς την αντιπολέτευση για να ασκηθεί, να μειωθεί η πόλωση, αλλά πώς θα γίνει αυτό αν δεν κάνει η κυβέρνηση το βήμα αυτό για τη μείωση του ποσοστού του 10%. Να συμφωνήσω επίσης με τον συνάδελφο, ο Μπιόλες, είναι ε, δύσκολη αυτή η ημερομηνία και καταλεκτική για την υποβολή των ε, τροπολογιών. Μπορούμε να το αναβάλουμε λίγο. Σας ευχαριστούμε. Για δύο λεπτά έχει το λόγο η κυρία Φλότρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ρία. Νομίζω πως όπως κάθε χρόνο πια μας παρουσιάζει ένα έγγραφο εργασίας πολύ τεκμηριωμένο, πολύ σοβαρό και πολύ εμπεριστατωμένο για το σύνολο των σημείων που θέλουμε να εξετάσουμε και είναι εξαιρετικά ε, ευχάριστο για μας του shadow, τους σκεώδεις, να μπορούμε να δουλέψουμε με αυτή τη βάση, την τόσο συμπαγή, την τόσο στέρεη. Στο πλαίσιο τώρα που σήμερα χαρακτηρίζει τη διαδικασία διαπραγματεύσεων και τις σχέσεις με την Τουρκία, δηλαδή ένα είδος κόπωσης αμοιβαία επικρατεί, θα πρέπει να μπορέσουμε με αυτή την έκθεση να στείλουμε μηνύματα πιο ξεκάθαρα, ακόμα πιο ξεκάθαρα και κάθετα μηνύματα που δίνοντας αυτή την έκθεση για ένα σύνολο σημείων ένα πιο, πιο, πιο μεγάλη έμφαση. Δηλαδή Καλύτερα να ξεκαθαρίσουμε τα φωτεινά και τα σκοτεινά σημεία, ώστε να χρησιμεύσει για την ενεργοποίηση της επικοινωνίας ανάμεσα στην ΕΕ και την Τουρκία και τους ε, Τούρκους ε, συναδέλφους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό νομίζω, λόγω του πλαισίου στο οποίο βρισκόμαστε. Για παράδειγμα, για την ελευθεροτυπία και την ελευθερία έκφρασης, που είναι ένα βασικό θεμέλιο ο κάθε δημοκρατική κοινωνία θα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο ξεκάθαροι, ακόμα πιο επικριτικοί. Η κατάσταση δεν είναι αποδεκτή και πρέπει να το πούμε όσο γίνεται πιο έντονα και να εκδηλώσουμε ακόμα περισσότερο την αντίρρησή μας, ακόμα περισσότερο τις ανησυχίες μας και τις απαιτήσει που έχουμε σε αυτό το θεμελιώδες ε, ζήτημα. Επίσης με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να υποστηρίξουμε με την διαδικασία μεταρρύθμισης συνταγματική μεταρρύθμιση, συγχωρείτε. Πάντοτε όμω σημειώνοντα, και γι' αυτό θα πρέπει νομίζω να επιμείνουμε, ότι δεν θα πρέπει να φυστούμε προσπαθειών πολιτικών ε, ε, πρωτοβουλειών και νομιμότητας για να ξυπνήσουμε τα κράτη-μέλη, την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Να στηρίξουμε νέες συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, αλλά ταυτόχρονα να καλέσουμε εξίσου ξεκάθαρα το Συμβούλιο να ανοίξει το κεφάλαιο 23-24 για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τη δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ναι, ναι, τελειώνω. Δεν θα μακρηγορήσω άλλο. Κατά τη γνώμη μου, για το Κυπριακό υπάρχει ένα αίτημα που δεν νομίζω ότι εντάσσεται στο πλαίσιο των ε, σημερινών διαπραγματεύσεων και εδώ νομίζω ότι μία εφαρμογή του πρωτοκόλλου θα πρέπει να υπογραμμιστεί. Αυτό το κάνετε. Μπορούμε επίσης να ζητήσουμε από την Ένωση να ενεργοποιήσει αυτόν τον κανονισμό, όπως έχει δεσμευτεί για το άμεσο εμπόριο με την Βόρεια Κύπρο. Ταυτόχρονα εγώ λοιπόν κάνω έκκληση για ενεργοποίηση του πολιτικού μηνύματος, δηλαδή να δώσουμε και να στείλουμε μηνύματα ώστε να ενεργοποιηθεί και πάλι ο διάλογος και οι διαπραγματεύσεις. Η κυρία Γιαννάκου για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τη συνάδελφό μας κυρία Όμεν για την επανάληψη της έκθεσής της, η οποία πραγματικά αποτυπώνει και την πρόοδο που έχει γίνει σε ορισμένους τομείς ε, και τα αρνητικά σημεία, όπως παραδείγματος χάρη είναι η μία αναγνώριση της Κύπρου. Πώς είναι δυνατόν μια χώρα υποψήφια να μην αναγνωρίζει τα κράτη-μέλη. Εκείνο που ήθελα να επισημάνω ε, στην κυρία Οούμενη είναι ότι δυστυχώς παρά το γεγονός ότι το Μάιο του 10 έγινε ένα high level meeting και δημιουργήθηκε μια ομάδα ανάμεσα σε υπουργού και τους Πρωθυπουργού, και ήρθε ο κύριος Ερντογάν στην Αθήνα με δέκα υπουργούς για τις σχέσεις καλής γειτονίας δεν υπάρχει ουσιαστική πρόοδο και οι υπερπτήσεις πάνω από το Αιγαίο σε λιγότερο από έξι μίλια από τα ελληνικά νησιά συνεχίζονται και το χειρότερο συνεχίζονται οι υπερπτήσεις πάνω από το έδαφος οπλισμένων βομβαρδιστικών ε, και θεωρώ ότι αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό για να περιληφθεί στην έκθεση. Είναι πρότασή μου προς την εισηγήτρια, η οποία κατά τα άλλα είναι εξαιρετική. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Γιαννάκο. Ο κύριος Χατζηγεωργίου, δύο λεπτά. Ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Νόουμε. Εμείς ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακολουθούμε με πολύ προσήλωση τι προσπάθειε που καταβάλει η τουρκική κοινωνία να εκδημοκρατιστεί, να προχωρήσει σε αλλαγέ δομών είτε στο Σύνταγμα είτε σε άλλε ψυχέ τη πολιτική και κοινωνική ζωή, γιατί θεωρούμε ότι αυτό θα είναι προ όφελο και τη Τουρκία και των χωρών που είναι γύρω από την Τουρκία αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θεωρούμε όμως ότι το συγκεκριμένο report της κυρίας Σόουμεν, το οποίο ε, αναλύει τα πράγματα προς σωστή κατεύθυνση πρέπει να εμπλουτιστεί με μερικά στοιχεία τα οποία είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά. Πρέπει καταρχήν όσον αφορά το Κυπριακό, κατά τη δική μας άποψη, να περιγραφεί ποια είναι η λύση που αναζητούμε. Η βάση της λύσης την οποία αναζητούμε για μας έχει σημασία γιατί γίνονται συνομιλίες και κανένας δεν πρέπει να έχει την ε, την ιδέα ή την σκέψη στο μυαλό του ότι αυτό το πράγμα μπορεί να αλλάξει. Πρέπει να γίνει μια αναφορά για την Αμόχωστο. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Αμόχωστος είναι μια πόλη που εδώ και 36 χρόνια κατοικείται από φίδια και ποντίκια. Αυτό δεν ευαισθητοποιεί τους Ευρωπαίους. Μια πόλη η οποία καταραίει μέσα σε ερήπια. Μια ευρωπαϊκή πόλη με μια ιστορία τόσο συνδεδεμένη με τον ευρωπαϊκό χώρο όσο πολύ λίγες ε, πόλεις της ε, περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Νομίζω ότι το report πρέπει να συμπεριλάβει την ανάγκη άμεσης επιστροφής μιας πόλης ακατοίκητης από ανθρώπους, επαναλαμβάνω εδώ και 36 χρόνια. Δεν έχει σημασία ποιοι είναι οι κάτοικοι, οι ή οι Έχει σημασία ότι είναι μια πόλη εκεί ε, αδιανή. Κλείνω με το εξής. Η Τουρκία πρέπει να επιτρέψει τις υπερπτήσεις κυπριακών αεροσκαφών πάνω από το έδαφος της. Νομίζω είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που δεν επιτρέπει πτήσεις άλλων αεροσκαφών πάνω από το έδαφος της. Ευχαριστώ. Ε, Ο κύριος Σαλαβράκος, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, Θέλω να συγχαρώ εν πρώτη στην κυρία Όμεν Ρόιτεν, διότι έχει συντάξει μια έκθεση απόλυτα ισορροπημένη. Έχει επισημάνει ακριβώς τα σημεία στα οποία η Τουρκία έχει κάνει βήματα μπρος και έχει υπογραμμίσει τα σημεία στα οποία η Τουρκία εξακολουθεί να παραμένει στο κακό της παρελθόν. Ε, ξέρετε, παρακολουθώ το θέμα εδώ και πολλά χρόνια και διαπιστώνω από πλευρά μεν της κυβερνήσεως Ερντογάν μια προσπάθεια να κάνει πέντε βήματα εμπρός, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπω ότι και το διαπιστώνουμε αυτό κάθε μέρα ότι υπάρχουν πολλά κέντρα εξουσίας σε αυτή τη μεγάλη χώρα τα οποία έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση η οποία είναι αλλοπρόσωλη. Και το λέω αυτό για τον εξή λόγο. Την ώρα που η επίσημη κυβέρνηση Ερντογάν την χείρα φιλίας προς τις γειτονικές χώρες και λέει δια το στόμα του του Υπουργού Εξωτερικών της του κ. Νταβούτογλου ότι έχει μηδενικά προβλήματα στην περιοχή την ίδια ώρα κάνει παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου της Ελλάδος με μαχητικά αεροσκάφη οπλισμένα. Ήδη χθε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας και το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδος εξέδωσε ανακοίνωση ότι 18 τουρκικά αεροσκάφη εισήλθαν στο Φύρ Αθηνών χωρίς να καταθέσουν σχέδιο και κατεγράφησαν 14 παραβιάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο Φύρ Αθηνών που εξελίχθηκαν σε 13 παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου μεταξύ των νήσων Λέσβου και Χίου. Πιστεύω ότι δεν προάγει ούτε το κλίμα ενώσεως της χώρας αυτής με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ούτε το κλίμα της καλής γειτονίας προς τα γειτονικά της κράτη η όλη συμπεριφορά της Τουρκίας. Από την άλλη πλευρά, συμμερίζομαι το γεγονός ότι έχουν γίνει ορισμένες πρόσφατες συνταγματικές μεταρρυθμίσεις που δείχνουν ότι σε επίπεδο λαϊκής αποδοχής ο Ερντογάν απολαμβάνει μια μείζωνος εμπιστοσύνης. Ελπίζω την εμπιστοσύνη αυτή την οποία κατά από τα αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων φαίνεται να την αξιοποιήσει διότι μέχρι τώρα δεν φαίνεται ορατό ότι έχει αξιοποιήσει αυτή την αποδοχή τη λαϊκή και επιτρέπει στους ιέρακες της Τουρκίας να δημιουργούν αυτές τις καταστάσεις. Πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι η Τουρκία πρέπει να ζήσει στον κόσμο και ο κόσμος είναι έτοιμος να αποδεχθεί την Τουρκία να ζήσει με αυτόν. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να το, συνειδητοποιήσει η Τουρκία η οποία συμπεριφέρεται ως να μην χαμπαρίζει κανέναν άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Σαλαβράκο. Ο κύριος Χάουιτ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Μαναγάιτεν. Υπάρχει ε, βρήκατε συνένεση. Εγώ συν... Ε, σας συγχαίρω για τη διάφορα που έχετε γράψει εδώ. Ε, αλλά θα πρέπει όντως να μιλήσουμε για την αποτυχία, να ανοίξει το κεφάλαιο για την αποτυχία, ε, για τον ανταγωνισμό, συγγνώμη. Επίσης έχουμε την ολομέλη μετά από τη Σύνοδο του Συμβουλίου και άρα θα πρέπει να ενημερώσουμε τη διατύπωση και να σκεφτούμε και την δράση της κυρίας Άστον όσον αφορά τη στρατηγική συνεργασία. Επίσης να μιλήσουμε για τα όσα είπε ο κύριος Φούλη για το συνταγματικό δημοψήφισμα ανεξαρτησία ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος, ελευθεροτυπία, συμφωνώ με τα όσα λέει η συγγήτρια αλλά υπάρχει θέμα εφαρμογής το οποίο θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε ε, ε, οδηγίες προς τους εισαγγελείς αυτά που είπαμε πέρυσι έπειτα δεν, υπα... δεν είναι σωστό να λέμε πως δεν υπήρξε πρόοδος για την ανεξή θρησκεία αλλά συμφωνώ για τα όσα λέει για συγκεκριμένες θρησκευτικέ κοινότητες στην παράγραφο 23 νομίζω θα πρέπει να αναφέρουμε ότι υπήρξε αύξηση για τις δολοφονίες παλιότερα φαίνεται ότι καλύπτονταν όντως δεν θα πρέπει να δείξουμε καμία ανοχή στην παράγραφο 28 να αναφερθούμε στην ανάπτυξη της Ανατολής στην παράγραφο 39 να μιλήσουμε για καταδικάζει και όχι απλώς ε, λυπάται. Όσον αφορά την Κύπρο, στην ομάδα μου εν μέρη επιτύχαμε με τους Κύπριους ε, συναδέλφους ε, στη συζήτησή μας να βρούμε συνένεση και να διατηρήσουμε δίκαιη και επικοδομητική διατύπωση. Θα προσπαθήσουμε να το ξανακάνουμε και φέτος με τον συνάδελφο κύριο Μπιόλος και θα ζητήσω από την κυρία ο να το κάνει αυτό εξ ονόματος ολόκληρης Επιτροπής και πάλι το διπλόρ θα πρέπει να τα αλλάξουμε στο regret και η άμεση απόσυρση των, ομα... στατευμάτων πέρσι είχε αντιπαραγωγικό αποτέλεσμα και θα πρέπει διαφορετικό να το διατυπώσουμε για να γίνει αποστατικοποίηση. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να καθυστερήσουμε την υποβολή προθεσμιών γιατί χρειάζεται χρόνος εντός των ομάδων μας αλλά και εκτός του Κοινοβουλίου για να συντάξουμε τροπολογίες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Χάουιτ. Το κύριο Κασουλίδης για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Όμεν που μας παρουσίασε μία ισορροπημένη και αντικειμενική έκθεση και μάλιστα υψηλών προδιαγραφών, όπως είπε και ο κύριος Λάμστορφ. Τα θέματα της έκθεσης είναι καταρχήν τα κριτήρια της Κοπενχάγης, οπότε είναι ομόφωνη η ανησυχία μας ό,τι αφορά την ανεξιθρησκεία και την ελευθεροτυπία ή η ελευθερία έκφρασης ή ο σεβασμός των θρησκευτικών μειονοτήτων. Σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, έχω κάποιες ανησυχίες για τη νέα πολιτική της Τουρκίας απέναντι στο Ιράν και το Ισραήλ. Για την Αρμενία τίποτα δεν έχει γίνει. Δεν ήταν ουσιαστική η πρόοδος που έγινε, ήταν εικονική. Θα ήθελα επίσης να πω εδώ σε όλους ότι το πρόβλημα που φορά το άνοιγμα των διαπραγματευτικών κεφαλαίων με την Τουρκία δείχνει την ε, ε, αιμονή της, του, του ανοίγματο ε, του πρωτοκόλλου της Άγκυρας και η Τουρκία έχει παγώσει 8 και άλλα κεφάλαια. Αυτό δεν έχουν μείνει κεφάλαια που μπορούν να ανοίξουν. Προσοχή λοιπόν. Προσοχή με τα μηνύματα που δίνουμε. Θέλουμε να είμαστε λιγότερο επικριτικοί απέναντι στη Τουρκία. Να είμαστε μάλλον αυστηροί, επικριτικοί σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ως αντάλλαγμα να το εξισορροπήσουμε με την Κύπρο, έτσι θα βοηθήσουμε την, ε, ε, διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων. Ας το ξανασκεφτούμε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κύριε Κασουλίδη. Πριν να δώσω το λόγο στον επόμενο μιλητή, θέλω να σα πω ότι μετά από διαβουλεύσει με τη Γραμματεία, ότι μπορούμε να καθυστερήσουμε για μια εβδομάδα την υποβολή των τροπολογιών. Αντί για 10 ε, του μηνό, να είναι 18 του μηνό η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Έτσι ώστε να σας ικανοποιήσουμε. Ο κύριος Μαυρονικόλας, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και με τη σειρά μου και εγώ να δώσω συγχαρητήρια στην εισηγήτρια για την έκθεσή της. Θα ήθελα να αναφερθώ αποκλειστικά σε ένα σημείο σε ό,τι αφορά το κυπριακό πρόβλημα. Μπορεί το κυπριακό πρόβλημα να μην είναι λυμένο σήμερα, η δυνατότητα και η πιθανότητα να το λύσουμε στο μέλλον εξαρτάται αποκλειστικά από την δυνατότητά μας να σταματήσουμε την Τουρκία από το να συνεχίζει τον επικισμό των κατεχομένων. Πρέπει η Τουρκία να σταματήσει τη δημογραφική αλλαγή στα κατεχόμενα για να δώσει προοπτική και στο εγγύς και στο απότερο μέλλον για λύση του κυπριακού προβλήματος το αντίθετο θα συμβεί εάν με, εάν με τον συνεχιζόμενο επικισμό βρεθούμε ξαφνικά να προσπαθούμε να λύσουμε το κυπριακό πρόβλημα ομιλώντας με Τούρκους υπήκους και ήδη η πλειοψηφία στα κατεχόμενα είναι Τούρκοι υπήκοοι και όχι η τουρκοκυπριακή κοινότητα. Το αναφέρνω αυτό κυρία εισηγήτρια με την έννοια ότι στην περσινή χρονιά υπήρχε ένα amendment, μια τροπολογία η οποία μιλούσε για αυτό το θέμα προτινόμενη από τον κύριο Σβόποτα. Θα ήταν ευχής έργων αν μπορούσε αυτό το θέμα να αναφερθεί στην εισήγησή σας. Τη διαβάζω στα αγγλικά. Calls on... Ζητά από την Τουρκία και τις τουρκο... τουρκοκυπριακές αρχές να απόσχουν από οποιαδήποτε δραστηριότητα επικισμού Τούρκων στο νησί, γιατί αυτό θα εξακολουθεί να τροποποιεί τη δημογραφική ισορροπία και μειώνει την δυνατότητα εφαρμογή ενός κοινού, ενός νέου κράτου με βάση το κοινό παρελθόν. στην εισήγησή Ευχαριστώ Ο κύριος Πέτερλε για δύο λεπτά. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ την κυρία Όμαν την εισηγήτρια. Είναι πολύ καλή η έκθεση και χαίρομαι ιδιαίτερα είναι πάρα πολύ εύγλωτος ο τρόπος που αναφέρει τα γεγονότα. Τρία βασικά μηνύματα. Καταρχάς, η αναγνώριση της πρόοδου. Πολλά πράγματα πριν από κάποια χρόνια ήταν αδιανόητα. Αλλά ξέρουμε ότι σήμερα έχουμε πολλές νέες εξελέξεις. Φυσικά αναμένουμε να εφαρμοστούν και όλα αυτά. Κατά δεύτερον, περιμένουμε να συνεχιστούν δυναμικά οι μεταρρυθμίσεις και κατά τρίτον θα πρέπει να εξετάσουμε τα βασικά προβλήματα σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις για την προσχώρηση και φυσικά το Κυπριακό έχει ε, μπει στο προσκήνιο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό η Τουρκία περιμένει από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιες συγκεκριμένες δράσεις, πράξεις. Και αυτό μας βρίσκει κάπως αντίθετους. Σύμφωνο ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την διαδικασία αυτή και να υποστηρίξουμε πλήρως τις πράξεις εκείνες, τις δράσεις εκείνες που θα καταλήξουν σε μια οριστική λύση. Και σε ό,τι αφορά τις ε, συνταγματικές ε, αναθεωρήσεις. Γιατί αν υπάρξει μεγαλύτερη πόλωση δεν θα συνεχιστούν οι αλλαγές. Τέλος, ε, τελευταία μάλλον, ο αριθμός των κοινοβουλευτικών επαφών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ε, τουρκικών κομμάτων και της αντιπολίτευσης μάλιστα ε, αυξήθηκαν. Νομίζω ότι κατανοούμε καλύτερα πλέον την κατάσταση και αυτή η κοινοβουλευτική διάσταση θα πρέπει να εμαθυνθεί. Και τέλος η οικονομία αναφέρθηκε στην έκθεση της κυρίας Όμαν Ράιτον θεωρώ ότι δεν είναι μόνο θέμα ευελιξίας της τουρκικής οικονομίας. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε περαιτέρω τα τουρκικά επιτεύγματα και θα ήθελα να τα δω και στην Ευρώπη. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που η τουρκική οικονομία και οι εκπρόσωποι της έχουν καλές επαφές με τον οίκο μας. Ευχαριστώ κύριε Πέτερλε. Ο κύριος Φόμποτα, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάποιες παρατηρήσεις. Νομίζω ότι με κάποιο τρόπο θα πρέπει να αναφέρουμε κάτι το οποίο συνεπάγεται και το άνοιγμα των κεφαλαίων δεν είναι μόνο το κυπριακό και συμφωνώ με αυτά που είπε ο συνάδελφος Μαυρονικόλα σε ό,τι αφορά την ε, πολιτική του επικισμού και το πρωτόκολλο της Άγκυρας και η Τουρκία δεν είναι έτοιμη και κάποια κρατημέλη δεν είναι έτοιμα ακόμα. Να το πούμε και αυτό, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που αποτρέπουν την εξέλιξη κατά δεύτερον. Γι' αυτό που είπε η συνάδελφος Όμεν Ρόιτεν, μάλλον ε, αυτά που αναφέρει ό,τι αφορά την ανταπαράθεση στο εσωτερικό του πολιτικού φάσματος ε, στην Τουρκία, συμφωνώ. Θα ήθελα να αναφέρω ότι ο Ερντογάν μετά το δημοψήφισμα τόνισε ότι ήταν σφάλμα να μην υπάρξει ευρύτερη βάση και αυτή την υπόσχεση κατά πόσο θα την θυμηθεί και κατά πόσο θα αποπειραθεί να προσεγγίσει τα άλλα ε, κόμματα και την αντιπολίτευση. Δεν ξέρω, δυστυχώς ε, και στο εσωτερικό της αντιπολίτευσης υπάρχουν διχασμένες απόψεις και επίσης για αυτό που είπατε για την κοινωνική διάσταση συμφωνώ επίσης για την Αρμενία. Θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να ξεκινήσει νέος ε, διάλογος μεταξύ Αρμενίας και Τουρκίας θα πρέπει να επικυρωθούν τα πρωτόκολλα. Ξέρουμε ότι συνδέονται και με τα θέματα του Αζερβαϊτζάν και του Αγκόρνο Καραμπάχ, αλλά είναι ε, απαραίτητο να υπάρξει ένας νέος διάλογος για το θέμα το κουρδικό τώρα και εδώ συμφωνώ ότι έχουν συμβεί πολύ περιορισμένα πράγματα. Υπάρχει θέληση, έχουν γίνει κάποια δηλαδήματα, αλλά θα πρέπει να υπάρξει τόλμη για να γίνουν περαιτέρω βήματα παρά τις τρομοκρατικές ε, επιθέσεις. Θα πρέπει η Τουρκία να βρει την τόλμη για να προχωρήσει. Θεωρώ ότι συνολικά είναι πολύ ισορροπημένη η έκθεση για το θέμα της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια μεγάλη ευκαιρία για την εξωτερική πολιτική, αλλά θα πρέπει να γίνει αυτό ε, ε, σε συμφωνία, σε αρμονία με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι ανεξάρτητα από αυτή. Είναι πολύ σημαντική η πτυχή αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σβόμποντα. Η κυρία Μποσκούρτου. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε και καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ρία Όμεν για την προσοχή που δίνει στο θέμα των ε, δικαιωμάτων των γυναικών στην έκθεση. Είναι πάρα πολύ σημαντικά σημεία αυτά για τα οποία είχα ζητήσει να δοθεί προσοχή. Χαίρομαι που αναφέρεται το θέμα των ποσοστώσεων επιτέλους. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν Ρία. Δεύτερο ζήτημα η έκθεση φυσικά μου θυμίζει πολλά πράγματα ασφαλώ σε σχέση με το παρελθόν. Μου προκαλεί ένα déjà vu. Αλλά μου λείπουν και κάποια στοιχεία. Για παράδειγμα, προσοχή στην πρόσφατη κατάσταση σε ό,τι αφορά το θέμα των, της μαντήλας στα πανεπιστήμια. Δεν επανέρχεται. Είναι σημαντικό όμως για την Τουρκία. Τα δικαιώματα για τους ομοφιλόφιλους και η παράγραφος για την Συμφωνία Εταιρικής Σχέσεως και θέματα για τις θεωρήσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά και υπάρχουν ε, περιπτώσεις που καταδεικνύουν ότι υπάρχουν ζητήματα σχετικά με τα ε, ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε υποσχεθεί σχετικέ έρευνε, τι θα σημαίνει αυτό για τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά δεν επανέρχονται στην έκθεση. Ελπίζω λοιπόν να δοθεί προσοχή. Τελευταίο σημείο που θέλω να θίξω. Είναι σαφέ ότι μας τελειώνουν τα κεφάλαια προς διαπραγμάτευση. Ασφαλώς αυτό εν μέρη το προκαλεί η ίδια η Τουρκία, αλλά και κατά μεγάλο μέρος το προκαλούν και τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επειδή μας τελειώνουν τα κεφάλαια, νομίζω ότι χρειάζεται πλέον μια στρατηγική για να δούμε τι μπορεί να γίνει για να συνεχίσουν, να, να ξαναξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Αυτά λοιπόν ήταν τα στοιχεία που ήθελα να αναφέρω και να ευχαριστήσω εκ νέου την Ρία για τις προσπάθειες που έκανε. Σα ευχαριστώ. Κόβατσεφ, δύο λεφτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Ρία Όμεν για την πολύ ισορροπημένη της έκθεση. Τα περισσότερα της σημεία είναι ισορροπημένα και σωστά. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο σημεία. Το 36 που συνδυάζεται το θέμα της έναρξης ε, του κεφαλαίου για την ενέργεια με την ε, διακυβερνητική συμφωνία για το Ναμπούκο. Δεν τελειώνω όμως αυτά τα θέματα. Θέλουμε να υποστηρίξουμε το σχέδιο Ναμπούκο η Βουλγαρία, η Αυστρία, η Ρουμανία και η Ουγγαρία. Όλες οι χώρες που συμμετέχουν είναι έτοιμες να ε, υπογράψουν το σχέδιο στήριξης της συμφωνίας Ναμπούκο. Αλλά φαίνεται ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί την προθυμία των χωρών για υπογραφή της συμφωνίας ε, για να πιέσει για το άνοιγμα του κεφαλαίου, του διαπραγματικού κεφαλαίου για την ενέργεια. Δεν θέλω να πιέζει με τέτοιο τρόπο η Τουρκία την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία για να ανοίγει ένα κεφάλαιο. Δεν είμαστε κατά του ανοίγματο του κεφαλαίου για την ενέργεια, αλλά όχι υπό τον όρο της ή σε συσχετισμό με την ε, συμφωνία αυτή του στη, τη στήριξη για τον Ναμπούκο. Όχι να μας δίνει τελεσίγραφο δηλαδή η Τουρκία ότι αν δεν ανοίξετε το κεφάλαιο για την ενέργεια εμεί δεν θα υπογράψουμε το σχέδιο στήριξης ε, του Ναμπούκο. Να μην γίνεται συσχετισμό. Σε ό,τι αφορά την επικύρωση των πρωτοκόλων για την Αρμενία, ήταν σαφέ από την υπογραφή ε, του πρωτοκόλου στην Ελβετία ότι δεν ήταν προποθέσει. Τώρα και ο σχετισμός αυτών των πρωτοκόλων με, τις παγωμένες συγκρούσεις ε, στον Αγκόρνο Καραμπά και το Σερβαϊτζάν κατά τη γνώμη μου δεν συνάδει με την προσπάθεια δημιουργίας εμπιστοσύνης ε, στην Τουρκία μεταξύ των γειτονικών τους χωρών. Σίγουρα μία συμφωνία θα πρέπει να στηρίζεται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη και αμοιβαία εμπιστοσύνη σημαίνει ε, σεβασμός των ηλυμένων αποφάσεων και των πρωτοκόλων που έχουμε υπογράψει. Κύριε Μπρέπολης, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω στην κυρία Όμουν Ράιτον ότι συμφωνώ με τα κριτικά σημεία που αναφέρει στην έκθεσή της σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, το δημοκρατικό άνοιγμα, η οποία, το οποίο ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί συγκεκριμένα το δημοψήφισμα επίσης. Έχει έρθει λοιπόν η ώρα να εφαρμοστούν αυτά και συμφωνώ σε ό,τι αφορά θέματα τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν συγκεκριμένα. Να μιλήσω όμως συγκεκριμένα για τις παραγράφους για το κουρδικό. Θα πρέπει θεωρώ να γίνουν πιο ε, να γίνει πιο οξία η διατύπωση και θα κάνω σίγουρα σχετικές τροπολογίες γιατί δεν αναφέρεται για παράδειγμα η διαδικασία η οποία ε, γίνεται αυτή τη στιγμή στο Μπακύρ κατά 150 ε, δημοκρατικά εκλεγμένων πολιτικών, Κούρδων και ακτιβιστών. Επίσης ότι ε, αγνοούνται συστηματικά τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος και δεν αναφέρονται λοιπόν όλα αυτά τα ζητήματα και η διαδικασία, η αγωγή κατά του Ρόσκοβη στην Δανία και στο Βέλγιο και σε άλλες χώρες. Ε. Επίσης ε, ασκείται κριτική για το ΠΚΚ, αλλά δεν αναφέρεται τίποτα για παράδειγμα για την ανακοχή. Με άλλα λόγια, θεωρώ ότι θα πρέπει να αναφέρουμε με σαφήνεια ότι η τουρκική κυβέρνηση θα πρέπει να ξεκινήσει διάλογο, διάλογο με Κούρδους εκπροσώπους για να καταλήξουν σε συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία θα οδηγήσουν στη συμπερίληψη και στο σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των Τουρκών πολιτών στην Τουρκία. Η κυρία Γκόμες για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τη συνάδελφο Ρία Όμεν Ρόιτεν για την ισορροπημένη, επικοδομητική και αντικειμενική της έκθεση. Συμμερίζομαι την άποψη εκείνων που είπαν ότι το θέμα του ανοίγματο κεφαλαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι σημαντικό και με απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα της ελευθεροτυπίας και της ελευθερίας έκφρασης. Ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των αποκαλύψεων της Wikileaks και του ρόλου που έπαιξε η Τουρκία στα, στο πρόγραμμα παράνομων παραδόσεων. Επίσης το θέμα των γυναικείων δικαιωμάτων, δικαιωμάτων γυναικών είναι νευραλγικό και είναι σημαντικό που αναφέρουμε και μία των ποσοστώσεων Καλό αυτό. Σε ό,τι αφορά την ε, πίεση για την ε, κύρωση του ICC, είναι πολύ σημαντικό και χαίρομαι που υπάρχει στην έκθεση. Για το θέμα της Κύπρου, νομίζω ότι είναι σημαντικό να καταλήξουμε σε συμφωνία μεταξύ μας και να βρούμε το σωστό τόνο και το ύφος για το μήνυμα που θα δώσουμε ως προς την Κύπρο. Το πιο σημαντικό πάντως είναι ότι το είναι συμφέρον τη Τουρκία, αλλά όχι μόνο τη Τουρκία, είναι θέμα συμφέροντο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει αυτό το σημείο να γίνεται αγκάθι και να εμποδίζει την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνα και το σχετισμό με τον ΝΑΤΟ εξαιτία των προβλημάτων που δημιουργούνται εξαιτία τη μη επίλυση του Κυπριακού. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι προτεραιότητα τρίτο σχόλιο. Ρία, μήπως θα μπορούσες να μας πεις δύο λόγια για την διαφθορά και την δωροδοκία, ιδιαίτερα στα θέματα τα οικονομικά και τα κοινωνικά, γιατί αυτό είναι το πρώτο πράγμα που α, βλέπει κάποιος όταν επισκέπτεται για πρώτη φορά την Τουρκία. Τεράστια φοροδιαφυγή. Και η διαφθορά ξεκινάει από τα χαμηλότερα κλιμάκια, οπότε αν υπάρχει τέτοια εκτεταμένη διαφορά στη βάση, τι θα γίνεται στην κορυφή. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό το θέμα της πάταξης διαφθοράς για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να το αμελούμε στη, στο κεφάλαιο με την Τουρκία. Ευχαριστώ και η κυρία Παπαδοπούλου για δύο λεπτά. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, να συγχαρώ την Ρία Όμεν για την έκθεσή της και συμφωνώ απόλυτα με τις ανησυχίες που εκφράζει για τις ελευθερίες, ε, σε ό,τι αφορά τα μέσα ενημέρωση στην Τουρκία, τα δημοκρατικά ελλείμματα τα οποία εξακολουθούν, εξακολουθούν να υπάρχουν σε θέματα δικαιωμάτων γυναικών, ε, στα βασανιστήρια, την καταπολέμηση τη διαφθορά, Θα πρέπει να είμαστε επικριτικοί έναντι τη Τουρκία, γιατί πρόκειται για μια χώρα υποψήφια, η οποία θα πρέπει να ε, σέβεται τι κοινέ ευρωπαϊκέ μα αξίε για να καταστεί μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. και δυστυχώ η Τουρκία δεν δείχνει οποιοδήποτε σεβασμό στην ε, Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές αξίες που προσβεύουμε. Δεν εφαρμόζει το πρόσθετο πρωτόκολλο και πρόκειται για μια υποχρέωση της Τουρκίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν αναγνωρίζει την Κύπρο. Και αυτό αποτελεί υποχρέωση της Τουρκίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, παραβιάζει τα ανθρώπινα και τα θρησκευτικά δικαιώματα των Ελληνοκυπρίων και έχει καταστρέψει την πολιτισμική μας κληρονομιά και πάνω από 500 εκκλησίες που συγκαταλέγονται στην κοινή ευρωπαϊκή μας ε, πολιτισμική ε, κληρονομιά. Επίσης θεωρώ ότι η κυρία Όμεν θα πρέπει να αναφέρεται την αμόχωστο στην έκθεσή σας και στην ανάγκη προστασίας ε, της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου και να σταματήσουν οι καταστροφές αυτές. Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται στην έκθεση η παράνομη επικισμή γιατί αποτελεί παραβίαση των εκθέσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης και επίση να υπάρξει αναφορά στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αγνοούμενων και των οικογενειών των αγνοούμενων στην Κύπρο. Για τα άτομα αυτά στην Κύπρο που έχουν υποφέρει εθνοκαθάρσεις τα τελευταία 36 χρόνια και αγαπητοί συνάδελφοι είμαστε 20.000 ε, Κύπροι που ζούμε σε αυτά τα ε, χώρια, σε αυτά τα χωριά. Σήμερα είμαστε λιγότεροι από 300 των αριθμών. Οι εθνοκαθάρσεις συνεχίζουν στην ε, Κύπρο. Να σταματήσουμε λοιπόν την ε, Τουρκία για να μην συνεχίσει αυτές τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ε, ανθρωπίνων αξιών. Σας ευχαριστούμε κυρία Παπαδοπούλου. Κλείνουν οι παρεμβάσεις με την κυρία Θεοχάρου για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα με τη σειρά μου να συγχαρώ την Ρίτα Ριαόμεν για τον ξεκάθαρο πολιτικό λόγο που έχει αρθρώσει μέσα στην έκθεση της και να επισημάνω ότι έχει θέσει και την βάση λύσης του κυπριακού προβλήματος με τον πιο σωστό τρόπο από όσους έχουν δει μέχρι τώρα το φως της δημοσιότητας. Σας συγχαίρω κυρία Ομέν διότι έχετε μιλήσει για λύση του κυπριακού στη βάση των αρχών και των αξιών και των θεμελιωδών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν νομίζω ότι υπάρχει οποιοδήποτε εδώ μέσα ο οποίος θα μπορούσε να διαφωνήσει σε αυτή τη βάση. Εμείς θέλουμε σε αυτή τη βάση να λυθεί το κυπριακό χωρίς καμία απόκληση και νομίζω ότι κανείς δεν θα δεχόταν να ισχύσει για τους Κύπριους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτι λιγότερο από ό,τι ισχύει για την δικιά του την χώρα. Βεβαίως κάποιοι επιμένουν να μην σέβονται θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Επιτροπή Νομικών η οποία είπε ότι η νομική βάση του ε, λεγόμενου απευθείας εμπορίου με τις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου είναι λαθεμένη και να ζητούν να επανέλθει το ζήτημα του απευθείας εμπορίου. Η απόφαση του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου του 2004 μιλάει για επανένωση της Κύπρου και όχι για μόνιμο διχασμό. Και όταν την επικαλούνται θα πρέπει να το θυμούνται και να την έχουν διαβάσει καλά. Γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι η έκθεση της κυρίας Όμεν πρέπει να αποτελέσει τη βάση για την παραπέρα πορεία μας όσον αφορά την επίλυση του Κυπριακού και τον εκδημοκρατισμό της Τουρκίας. Σας ευχαριστώ. <clears throat> Ah, Μάλιστα. Μια ακόμα παρέμβαση. Ο κύριος Λάμστορφ διαδικαστικό για θέματα της οργάνωσης των εργασιών με η συνάδελφος ε, Μενρό ήταν υπέβαλε μια έκθεση για την Τουρκία και υπάρχουν σκιώδεις εισηγητές φλότρ, ε, ομπιόντ κτλ. και εγώ νομίζω καλό θα ήταν οι σκιώδεις εισηγητές που ασχολούνται με το θέμα της ε, έκθεσης της Τουρκίας να έχουν πιο πολύ χρόνο αγόρευσης από τους άλλους συναδέλφους οι οποίοι φυσικά τους εκτιμούμε ιδιαίτερα αλλά δεν είναι έκθεση για την Κύπρο δεν είναι και έκθεση για την επίλυση του Κυπριακού και καταλαβαίνω φυσικά πόσο αφορά αυτό τους συναδέλφους και πόσο ευαίσθητο είναι το θέμα, αλλά να πω και προς τους Τούρκους φίλους ότι μπορούν να υπολογίζουν ότι οι μεγάλες ομάδες ε, του Κοινοβουλίου θα πραγματευτούν την έκθεση αυτή ως έκθεση για την ε, Τουρκία, όχι για την έκθεση για το Κυπριακό και θα ήθελα λοιπόν αυτό να αποτυπώνεται και στο χρόνο αγόρευσης. Μάλιστα. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Χριστόφ Φιλιόρη, που είναι επικεφαλής της, του αρμόδιου τμήματος της Επιτροπής. Παρακαλώ, σας ακούμε με ενδιαφέρον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πω σύντομα πως αυτή η έκθεση σε αυτό το στάδιο εξετάζεται πολύ προσεκτικά από πλευράς της Κομισιόν ε, θα περιορίσω λοιπόν τις παρατηρήσεις μου στη ε, προβλήματα που αφορούν τα πολιτικά κριτήρια για να εκφράσω άμεσα την πολύ θετική εκτίμηση της Επιτροπής για την έκθεση της κυρίας Όμεν Ρόιτον, η οποία πάνω σε αυτά τα θέματα των πολιτικών κριτηρίων αντικατοπτρίζει πολύ καλά την ισχύουσα κατάσταση στην Τουρκία. Τα συμπεράσματα συμπεριλαμβάνουν και τα ε, συμπεράσματα της Κομισιόν ε, την ετήσια έκθεσή της για την Τουρκία που δημοσιεύθηκε ε, το περασμένο Νοέμβριο. Μόνο μία παρατήρηση όσον αφορά τη συνεργασία κατά του τρομοκρατία. Να θυμίσω πως κυρίω η Τουρκία ζήτησε τα τελευταία χρόνια τη συνεργασία με την Ευρώπη. Ε, ίσως όπως το κείμενο έχει διατυπωθεί αυτή τη στιγμή στην έκθεσή σας μπορούσε να αφήσει να νοηθεί ότι εμείς εμέσως επικρίνουμε την Τουρκία για έλλειψη συνεργασίας σε αυτό το τομέα. Ε, ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε την ε, διόρθωση του κειμένου για το συγκεκριμένο σημείο. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ωραία. Να δώσουμε στην εισηγήτρια Όμεν Ρόιτεν ε, το τελευταίο λόγο. Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, όλους τους συναδέλφους για τις πολύ θετικές παρατηρήσεις και την θετική υποδοχή της έκθεσης. Είμαι ευγνώμων, πρόεδρε, να κάνω μία παρατήρηση άτακτη. Ελπίζω αυτό να αποτυπωθεί και στον αριθμό των τροπολογιών που θα κατατεθούν. Τρίτη παρατήρηση και να ξεκινήσω με τον ε, κύριο Ομπόης, ο οποίος ξέρει ότι εδώ στο Κοινοβούλιο είναι διχασμένες οι γνώμες σε ό,τι αφορά την εισδοχή της Τουρκίας. Και ελπίζω φέτος να μπορέσετε να το σεβαστείτε γιατί προσπάθησα και στις αιτιολογικές σκέψεις να διευκρινίσω ποιε είναι οι απόψεις σε ό,τι αφορά τη μελλοντική εισδοχή της Τουρκίας. Ελπίζω λοιπόν τη διατύπωση την οποία αφι... Ε, βάλαμε να μπορέσουμε φέτος να την αφήσουμε ως έχει, γιατί αποτυπώνονται οι αλήθειες χωρίς να θίγεται κανείς. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι περαιτέρω πόλωση στη συζήτηση αυτή δεν θα ωφελήσει ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε την Τουρκία. Δεν θα ήθελα λοιπόν να γίνει αυτό. Αυτά λοιπόν, Πρόεδρε, τα λέω προς τον κύριο Όμπες. Επίσης, για τον άλλο σκιώδη συγητή, τον συνάδελφο Χόουιτ, που ανέφερε κάποια στοιχεία και είπε ότι θα έπρεπε ίσως να τροποποιηθούν, να απαντήσω σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο ανταγωνισμού. Έχω την αίσθηση ότι για κάποια κεφάλαια και θα μπορέσει να μας το εξηγήσει, να σας το εξηγήσει καλύτερα ο εκπρόσωπος της Κομισιόν ότι έχει καθυστερήσει υπερβολικά η Τουρκία ή σε τελευταία στιγμή, τελευταία στιγμή υποβάλλει τα σχετικά σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό να σας πω ότι σε κάθε περίπτωση δεν φταίει η Ευρώπη. Έχω την αίσθηση ότι ακόμα δεν είναι έτοιμη η Τουρκία. Πρόεδρε, ο συνάδελφος Χάουετ έκανε και άλλες παρατηρήσεις σε ό,τι αφορά και τα εγκλήματα τιμής. Κοιτάξτε, δεν τα έχω μετρήσει, αλλά τα αριθμητικά στοιχεία που αναφέρω και τα περιστατικά που αναφέρω είναι αληθινά. Να είστε σίγουροι. Αυτό σημαίνει ότι από κάπου τα έχω βρει. Τα σωστά αυτά. Τα έχω βρει συγκεκριμένα τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ελπίζω λοιπόν να μην χρειαστεί να αλλάξουμε οτιδήποτε εδώ και δεν συμφωνώ επίσης σε ό,τι αφορά τις προτάσεις, σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, να πούμε regrets αντί για deplore. Όχι, δεν είμαι υπέρ πρόεδρο της πρότασης αυτής και γιατί, γιατί υπάρχουν φυσικά κάποιε κάποιες ε, Λέμε ότι καλό είναι ότι η Τουρκία έχει πραγματική εξωτερική πολιτική και ασχολείται ιδιαίτερα με αυτήν, αλλά αφετέρου φαίνεται ότι αποκλίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητώ λοιπόν από την ε, Τουρκία αλλά και από την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο να εργαστούν σκληρότερα προς την κατεύθυνση της σύγκλησης. Δεν αναφέρεται αυτό ρητά, αλλά ο τρόπος κατά τον οποίο μιλάει η έκθεση για το Ιράν και για το Συμβούλιο Ασφαλής κτλ. Κοιτάξτε, δεν πιστεύω ότι αυτό είναι απλά απογοητευτικό. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη διατύπωση επέλεξα. Να πάω στον κύριο Λάμστορτ τώρα, Αλεξάνδερ. Και εμένα δεν με ικανοποιεί η μη συμπερίληψη ε, του θέματος του ορίου του 10% και προσπαθώ να τους καλέσω να κάνουν κάτι προς την κατεύθυνση αυτή. Και θα πρέπει να ξέρεις ε, επίσης ότι δεν είναι μόνο τα μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης, το ΑΚ, αλλά και το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης έχει συμφέροντα σε ό,τι αφορά το 10% γιατί αυτοί είναι τελικά που ωφελούνται. Να το έχουμε υπόψη αυτό. Για την ελευθερία του τύπου το έθεσα πιο έντονα και έγιναν σχετικές συνομιλίες τον τελευταίο καιρό ως προς το θέμα αυτό. Ελπίζω λοιπόν να σας ικανοποιεί πλέον η διατύπωση. Πρόεδρε, ξεκίνησε μετά η κυρία Φλότρ λέγοντας, κάνοντας κάποιες παρατηρήσεις οι οποίες ε, ακολουθήθηκαν και από παρατηρήσεις του Αλεξάνδρου για το θέμα της Κύπρου. Διαπιστώνω ότι όλοι οι συνάδελφοι βρίσκονται εδώ, όλοι οι Κύπροι συνάδελφοι βρίσκονται παρόντες σήμερα εδώ και αυτό είναι καλό γιατί τους συμπαθώ ιδιαίτερα και τους γνωρίζω καλά. Αλλά θα ήθελα επίσης να πω, να πω το εξή. Εδώ ασχολούμαι με τη συγγραφή μιας έκθεσης για την Τουρκία. Και αν θέλουμε να επιλύσουμε το Κυπριακό, ε, θα βοηθηθεί η Τουρκία, θα βοηθηθεί η Ευρώπη. Αλλά βασικά είναι οι δύο κοινότητε στην ίσο που θα πρέπει να το κάνουν αυτό. Οι δύο κοινότητε στο νησί θα πρέπει να το κάνουν αυτό. Και αν θεωρείτε, και σα το έχω πει και κατηδίαν σε όλου, αν θεωρείτε ότι όλα όσα γράφω, και δεν ισχύει αυτό μόνο για την Κύπρο, αλλά και για άλλα κεφάλαια, όλα λοιπόν τα οποία έχω γράψει σε προηγούμενες θητείες και σε προηγούμενες ε, περιόδους, Κάθε χρόνο προσθέτω νέα στοιχεία και προσπαθώ σε κάποια χρόνια, ελπίζω να έχει επιληφθεί το θέμα, ελπίζω να έχουμε πιο πολύ Κύπρο από οτι, οτιδήποτε άλλο. Και σας το λέω, αν η κυρία Φλότρ ε, καταθέσει ως τροπολογία για τα θέματα άμεσου εμπορίου, ε, κατευθείαν εμπορίου, direct trade, αν ο κύριος Χάουιτ θέλει να αφαιρέσει θέματα σε ό,τι αφορά τα κατοχικά στρατεύματα και εδώ θέλετε να οξύνουμε την κατάσταση αναφέροντας την αμόχωστο και τίποτα άλλα, ε, θα είναι πάρα πολύ ωραία η έκθεση. Θα σπάσουμε ένα στο κεφάλι του άλλου, γιατί είναι πάρα πολύ διχασμένες οι απόψεις. Άρα, κατεπηγόντως, κατεπηγόντως τονίζω, σας καλώ όλους σας στο κεφάλαιο αυτό να αποδεχτείτε αυτά που έχω γράψει. Έχουμε αρκετά θέματα αναφέρει ως προς την Κύπρο. Έχουμε αναφέρει αρκετά συναισθηματικά ζητήματα ως προς την Κύπρο και στο θέμα των αγνοουμένων της πρόσβασης στις στρατιωτικές ζώνες που έχουν συμβεί μετά από εκθέσεις. Τα έχω συμπεριλάβει. Πάντα, σε κάθε περίπτωση τα έχω συμπεριλάβει. Σας παρακαλώ να είστε ικανοποιημένοι με αυτά που έχω γράψει. Μην καταθέσετε άλλες τροπολογίες και σας υπόσχομαι ότι δεν θα δεχτώ και τις τροπολογίες από την άλλη πλευρά. Ας αφήσουμε τα πράγματα ως έχουν γιατί αποτυπώνει ακριβώς αυτά που πρέπει να συμβούν. για να αξιοποιηθούν οι διαπραγματεύσεις προκειμένου να καταλήξουμε σε μια λύση γρήγορα. Πρόεδρε, ήθελα να αδειάσω την καρδιά μου και δεν θα ήθελα να ξεκινήσουμε όπως την προηγούμενη φορά μια τόσο ε, αντιφατική συζήτηση. Ελπίζω λοιπόν να είναι έτσι τα πράγματα. Πρόεδρε, να περάσω τώρα στον, στην αμήν. Το θέμα της ε, μαντήλας, κυρία Μποσκούρτ, δεν το ανέφερα, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι ευρωπαϊκό θέμα. Τελεία και παύλα. αυτά που είπες για τις θεωρήσεις. Θεωρώ ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το γνωρίζω το ζήτημα γιατί είναι ευρωπαϊκό ζήτημα. Πρόκειται για ένα πρόβλημα, μάλλον είναι ένα πρόβλημα το οποίο, θα πρέπει, το οποίο εμφανίζεται διμερώς σε ό,τι αφορά θέματα εκπαίδευσης. Ελπίζω να σε ικανοποιούν αυτά που ανέφερα για τον, για τον συνάδελφο Κόβατσεφ. Α, δεν είναι εδώ, έφυγε, ε, αλλά είπε, ανέφερε τον Αμπούκο. Πρέπει να το κοιτάξω. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοείται, αλλά δεν είχα την αίσθηση ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο σημείο αυτό. Η κυρία Μπρέπουλς ανέφερε τους Κούρδους. Δεν ξέρω τι θα έπρεπε να αναφέρω περαιτέρω, γιατί μας κατηγορεί συχνά η Τουρκία στην Ευρώπη ότι υποστηρίζουμε υπερβολικά το ΠΚΚ. Το ΠΚΚ είναι τρομοκρατική οργάνωση. Δεν θα ήθελα λοιπόν να ενισχυθεί και το ότι γίνονται συνομιλίες στην Τουρκία με τους Κούρδους είναι σαφές. Δεν ξέρω όμως αν θα έπρεπε να επισέλθουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Άννα σε ευχαριστώ που με υποστηρίζει σε ό,τι αφορά τη διαφθορά. Θα πρέπει να εξετάσουμε από κοινού κατά πόσον θα έπρεπε να συμπεριληφθεί κάτι άλλο. Πάντα συμπεριλάμβανα τέτοια στοιχεία, όχι όμω και αυτή τη φορά, γιατί δεν θέλουμε να επαναλαμβάνουμε τα ίδια συνέχεια, τα πάντα μάλλον συνέχεια. Αν θεωρείτε ότι είναι απολύτω απαραίτητο, να το κοιτάξουμε. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Φλόρη, παράγραφος 20 έχετε δίκιο. Το έχω ήδη αναφέρει ότι υπάρχει ένα λάθος. Πρέπει να αναφέρουμε ότι ενθαρρύνει την Τουρκία αλλά και την Ευρώπη να εντατικοποιήσουν την συνεργασία για τις ε, ενέργειες, τις τρομοκρατικές ενέργειες. Πρόεδρε, νομίζω ότι γρήγορα γρήγορα διέτρεξα όλα όσα ακούσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Check.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 Ήδη είπα ότι δίνουμε μία εβδομάδα παραπάνω για την υποβολή τροπολογιών σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που σας είχα πει αρχικά. Επαναλαμβάνω 18 Ιανουαρίου, 12 το μεσημέρι είναι τελική προθεσμία ενώ τα υπόλοιπα παραμένουν όσον αφορά την ψηφοφορία στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια. Περνάμε τώρα στο τελευταίο σημείο της ημερησίας διάταξης της σημερινής συνεδρίασης που αφορά την πρόταση ψηφίσματος για την σύναψη συμφωνία εταιρική σχέση και συνεργασία μέσα στην ΕΕ και των κρατών μελών τη με το Τουρκμενιστάν και τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνία εταιρική σχέση και συνεργασία με το Τουρκμενιστάν. Ένα σχέδιο σύσταση. Το λόγο έχει ο εισηγητή Νικολάη. Η εισηγήτρια, με συγχωρείτε, Νικολάη. Σα ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα έχουμε αρκετό χρόνο για να εξετάσουμε πλήρως αυτή την έκθεση. Είναι η δεύτερη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο. Εμείς σας ακούμε στο μικρόφωνο γιατί υπάρχει μια ψιλοβαβούρα αλλά στο μικρόφωνο σας ακούμε πολύ καλά. λοιπόν, έλεγα ότι ακόμα και αν έχει φασάρια στην αίθουσα εμείς στο μικρόφωνο σας το ακούμε πολύ καλά και μπορείτε να ε, συνεχίσετε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον, ε, τους σκιώδεις εισηγητές για τη συνεργασία τους στην εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Ε, είχαμε μια συνεδρίαση πριν λίγο καιρό και ε, συμφωνήσαμε για 13 συμβιβαστικέ τροπολογίε και για μια ολόκληρη σειρά τεχνικής, ε, τεχνικών τροπολογιών, οι οποίε ήταν ευπρόσδεκτε. Να κάνω μια διευκρίνηση. Η έκθεση αυτή ε, έχει μια προσέγγιση πολύ πιο επικριτική από ό,τι στην πρώτη της εκδοχή, αλλά περιέχει και μια αισιόδοξη πλευρά σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί η συμφωνία. Πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό και σημαντική συνεργασία με το Τουρκμενιστάν. Θα πρέπει εξίσου να τροποποιήσουμε τη στρατηγική μας, μια στρατηγική η οποία εδώ και 12 χρόνια αποτυγχάνει. Είναι μια στρατηγική απόλυτη απομόνωση του Τουρκμενιστάν στη διεθνή σκηνή. Θα ήθελα επίσης να επιμείνω για την ε, ε, συνεργασία μεταξύ μας που μας επέτρεψε να φτιάξουμε μηχανισμούς ελέγχου σε σχέση με αυτήν την συμφωνία και την εφαρμογή τους και με την έναρξη ισχύω της συμφωνίας της Λισαβόνας. Η θέση μας ε, μπορεί να είναι πιο δραστήρια σε σχέση με αυτές ε, τις συμφωνίες, δηλαδή αναθεώρηση για δύο χρόνια, συμφωνία για την Κεντρική Ευρώπη, Ασία με συγχωρείτε, Εκπρόσωπο του Συμβουλίου τη Κομισιόν και τη δική μα Κοινοβουλευτική Επιτροπή έχουν δραστηριοποιηθεί περισσότερο και έχει δημιουργηθεί και ένα μηχανισμό παρακολούθηση υπό την αιγίδα του ΥΠΑ εκπροσώπου μέσα στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Μια ολόκληρη σειρά λοιπόν νέων ιδεών που εισάγονται χάρη σε αυτή την έκθεση και κατά την άποψή μα αυτό μα επιτρέπει επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να δραστηριοποιηθεί πολύ περισσότερο. Μια ακόμα διευκρίνηση, χάρη στην έκθεση αυτή, προβλέπεται η συνεργασία ανάμεσα στα δύο Κοινοβούλια, το του Τουρκμενιστάν και του Ευρωπαϊκού. Είναι άρθρο είναι η παράγραφος 92 της έκθεσης. Εξάλλου πιστεύω ότι στο κοινοβουλευτικό πλαίσιο Δεδομένου ότι το Τουρκμενικό Κοινοβούλιο έχει γυναίκα πρόεδρο και το γεγονό επίση ότι η εκπροσώπηση των γυναικών είναι σημαντική στο Κοινοβούλιο του Τουρκμενιστάν είναι πάρα πολύ θετικό. Για την Κεντρική Ασία, δεν την περασμένη εβδομάδα, οι συνάδελφοι συμφώνησαν ότι πρέπει να συναυθεί μια συμφωνία συνεργασία. Εταιρική σχέση είναι μια συμφωνία απαραίτητη που θα πρέπει να μεριμνήσει για την ε, τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την ανάπτυξη. Αυτά όλα θεωρήθηκαν σημαντικά γιατί ε, για την ώρα έχουμε μόνο μια ενδιάμεση, μια προσωρινή συμφωνία που αφορά αποκλειστικά το εμπόριο. Νομίζω λοιπόν πως μόνο μια νέα συμφωνία θα μας επιτρέψει να ε, μπλακούμε περισσότερο στο Τουρκμενιστάν, ε, όχι μόνο από την άποψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και για τις οικονομικές σχέσεις. Θα ολοκληρώσω γιατί βλέπω ότι ο χρόνος πιέζει. Ελπίζουμε ότι στις 26 Ιανουαρίου, εφόσον ε, Η ψηφοφορία θα είναι ευνοϊκή και θα καταφέρουμε έτσι να αλλάξουμε την προσέγγιση μας στις διεθνείς σχέσεις και σε ιδιαίτερο στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ελπίζω λοιπόν πως θα περάσουμε από την παθητική ε, κριτική σε μια πολύ πιο δραστήρια εμπλοκή στις άλλες ώρες και πάλι μέσα στο σημερινό πλαίσιο με το Τουρκμενιστάν Πιστεύω πως η στρατηγική ισχύ που μπορούμε να έχουμε είναι ότι το γεγονό ότι το Τουρκμενιστάν θα μπορούσε να είναι μια οικονομική βιώσιμη ε, εταιρική σχέση. Είναι δύο στοιχεία τα οποία θα πρέπει να υπογραμμίσει το Ευρωκοινοβούλιο. Σα ευχαριστώ. Κυρία Νικολάη, το λόγο έχει ο κύριος Πέτερλε για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η συνάδελφος έκανε πολλές τροπολογίες και καταφέραμε με τον τρόπο αυτό να καθαρίσουμε το κείμενο προκειμένου να μην υπάρχουν ασυνέπειες και επαναλήψεις παρά τις ανησυχίες μας και παρά τις μεγάλες διαφορές θα θέλαμε να βρούμε μια βάση προκειμένου στο πλαίσιο αυτό να ενσωματώσουμε όλα εκείνα τα οποία πρέπει να συμβούν στο Τουρκμενιστάν. Αυτά από πλευράς μου. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Κιλ Νίλσεν για δύο λεπτά. Ε, Ευχαριστώ. Και εγώ θα συντάξω μια έκθεση για την Κεντρική Ασία τους επόμενους μήνες και θα προβώ σε μια αξιολόγηση της πρόοδου και στις πέντε χώρες ε, για τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Τουρκμενιστάν είναι μία από αυτές. Αυτό που με ε, εντυπωσιάζει σήμερα για το Τουρκμενιστάν είναι ότι μιλούμε για πρόοδο, αλλά θα ήθελα να σας επισημάνω δύο επιστολές, μία στα άλλη στην, ε, στο Γενικό Γραμματέα της ΟΑΣΕ στις 22 Νοεμβρίου και η δεύτερη επιστολή είναι ανοιχτή επιστολή. Έχουν υπογραφεί και δύο επιστολές από 19 ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτοί οι άνθρωποι και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις τους δεν μπόρεσαν να μεταβούν στο, στη διάσκεψη κορυφής ε, ε, στο Καζακστάν, όπου γινόταν ε, μία διάσκεψη κορυφή μεταξύ μη κυβερνητικών οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και μάλιστα απειλήθηκαν και στο Τουρκμενιστάν, αλλά και με την υποστήριξη του Καζακστάν δεν μπόρεσαν να μεταβούν σε αυτή τη ε, διάσκεψη κορυφής. Υπέστην ε, ε, και απειλές κατά της σωματικής τους ακαιρεότητας, μια κατάσταση εκφοβισμού και στις δύο επιστολές αναφέρεται ένα γενικό κλίμα στο Τουρκμενιστάν που κατά τη αξιολόγηση αυτών των μη κυβερνητικών οργανώσεων η περσινή χρονιά ήταν η πιο καταπιστική, η πιο ελεύθερη χρονιά προηγουμένω ότι αφορά τι επιθέσει κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καταστρατήγηση αυτών. Βλέπετε τι επιστολές, κάποιε μαρτυρίες με συγκλονιστικά συμβάντα. Αυτό είναι το γενικό κλίμα που επικρατούσε πέρυσι στο Τουρκμενιστάν, αλλά και φέτο ε, δεν καταδεικνύεται καμία ουσιαστική πρόοδος ότι αφορά τη βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή. Ευχαριστούμε κύριε Κιλ Νίλσεν. Το λόγο έχει ο Αντιπρόεδρος Πάσκου. Σας ευχαριστώ. Εδώ αντικαθιστώ τον κύριο Σίβιετ τον σκιώδη συγκητή μας, που μου ζήτησε να διαβάσω την ακόλουθη δήλωση που ουσιαστικά αντικατοπτρίζει τη θέση της ομάδας μας. Λέει λοιπόν ο κύριος Σίβιετ τη δήλωση αυτή. Είναι παλιό το δίλημα το κατά πόσο θα έχουμε ένα πλαίσιο συνεργασίας ε, με ατελείς δημοκρατίες ή με χώρες που έχουν αποτύχει παταγωδός ό,τι φορά την υλοποίηση των διεθνών προδιαγραφών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έτσι δεν μπορούν να επηρεάσουν θετικά την εσωτερική του κατάσταση ή να αρνηθούμε τέτοιου στενού δεσμού με τι χώρε αυτέ εξαιτία των αδυναμιών και των προβλημάτων που διαπιστώνουμε. Στην περίπτωση του Τουρκμενιστάν, διαπιστώσαμε κάποια πρόοδο ό,τι αφορά τι επιδόσει στα ανθρώπινα δικαιώματα. Βέβαια, ω προ τι μειονότητε ε, λίγο πιο σιγά, λέει ο πρόεδρο, πιο αργά παρακαλώ, γιατί δεν σα παρακολουθούν οι διερμηνεί και για του πολιτικού κρατουμένου. Έχει υπάρξει κάποια βελτίωση, αλλά πόρο απέχουμε από την ιδεώδη κατάσταση και θα πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερε προσπάθειε για να αντιμετωπιστούν αυτά τα ενισχυτικά προβλήματα. Οι συμβαστικέ πρωτοβουλίε που καταρτίστηκαν και συζητήθηκαν την εβδομάδα αυτή συνάδουν με τη θέση τη ε, ομάδα για την υπογραφή συμφωνία με το Τουρκμενιστάν η υπογραφή της Συμφωνίας Εταιρική σχέση βέβαια και συνεργασίας θα πρέπει να γίνεται υποαίρεση, υπό, υπό προϋποθέσεις και να περιλαμβάνει και την πιθανότητα αναστολής ε, της ε, υπογραφής αυτής της συμφωνίας με το Τουρκμενιστάν εφόσον δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του και δεν ανασυμβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υποστηρίζουμε τις συμβαστικές τροπολογίες. Η κυρία Χάουταλα, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγητριά μας για την πολύ αγαστή συνεργασία που είχαμε και την ανάλυση του αντικτύπου που θα έχει αυτή η Συμφωνία Εταιρική Σχέση και Συνεργασία στα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι περισσότερε συμβαστικέ τροπολογίε είναι εξαιρετικέ. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε κυρίω στο νέο μηχανισμό παρακολούθηση που εμπλέκει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτό ζητούν συμβαστικέ τροπολογίε. Είναι πάντως σωστό αυτά που επισήμαναν και οι συνάδελφοι. Και το μήνυμα της κυρίας Κιλ είναι σημαντικό. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ακόμη και σήμερα το καθεστώς του Τουρκμενιστάν είναι από τα πιο αυστηρά, αυταρχικά και καταπιστικά καθεστώτα του κόσμου. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη πριν συνενέσουμε για την υπογραφή της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας. Θα πρέπει να προβλέψουμε ένα μηχανισμό που να μας επιτρέπει να επαληθεύσουμε την βελτίωση της κατάστασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Τουρκμενιστάν. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να καταλήξουμε ε, στο συμπέρασμα αυτό ότι υπάρχει βελτίωση. Δεν μπορούμε ε, καλόπιστα και με το χέρι στην καρδιά αυτή τη στιγμή να πούμε ναι στη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας. Γι' αυτό και πολλοί συνάδελφοι είναι επιφυλακτικοί για το κατά πόσο θα πρέπει να δώσουμε το πράσινο φως στη συμφωνία ή όχι. Εμείς οι πράσινοι θεωρούμε ότι θα ήταν σκόπιμο να αφήσουμε την απόφαση αυτή για αργότερα, να περιμένουμε ένα χρόνο, να διαπιστώσουμε ότι το Τουρκμενιστάν δίνει τα σωστά μηνύματα, αυτό που περιμένουμε για τη βελτίωση. Γιατί αυτή τη στιγμή πραγματικά είναι αξιοθρύνητη η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή. Και ω προς το μηχανισμό παρακολούθησης φαίνεται ενδιαφέρουσα αυτή η καινοτομία που προτείνεται και επιμένω ότι ίσω θα είναι νευραλική σημασία για την ε, επίλυση του προβλήματος. Η διατύπωση όμως για τις πρώτες αυτέ είναι κάπως αόριστη. Θέλουμε ενίσχυση της διατύπωσης ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει τα εχέγγυα, να εξασφαλίσει τα εχέγγυα ότι όντω η Συμφωνία Εταιρική Σχέση και Συνεργασία θα βελτιώσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν θα αφήσει την κατάστασή του αμετάβλητη. Επίση, στη συμβαστική τροπολογία 2 που μιλάει για τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην παρακολούθηση συνδυασμό με την διετή αναθεώρηση τη ε, Συμφωνία Εταιρική Σχέση και Συνεργασία, η παρουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ενισχυθεί. Και κάτι περίεργο. Είχαμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 6 Φεβρουαρίου 1998 που, βλέπει, που προβάλλει το σχέδιο που από το παράρτημα 1 όμως ε, αφαιρείται το σημείο βοήθειας της κοινωνίας των πολιτών για, για το κράτος δικαίου. Ε, γιατί λείπει αυτό το σημείο, πού οφείλεται η διαφορά μεταξύ των δύο εκδοχών. Ευχαριστώ κύριος Γκζιμπ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την εισηγήτριά μας, αλλά και όλους ε, όσους κατέθεσαν τροπολογίες σε αυτή την έκθεση. Η έκθεση αυτή στην αρχή μας απογοήτευσε κάπως. Δεν ε, ε, ανταπεξερχόταν σε προσδοκίες μας ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και είχαμε κάνει πολλές στάσεις στο παρελθόν, αλλά δεν ε, ικανοποιήθηκαν δυστυχώς τα αιτήματά μας. Πάντως, ε, με τις ε, τροπολογίες βελτιώνεται η έκθεση και γίνεται πιο αντικειμενική. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να πιέσουμε το Τουρκμενιστάν. Θα πρέπει να επενέσουμε καταρχήν τη χώρα αυτή, να την εγκομιάσουμε για τα επιτεύγματά της, αλλά να μην περιοριστούμε σε κάποιες εικονικές πρόοδους. Θα πρέπει να είναι όντως γνήσια η πρόοδος που επιτέλεσε αυτή η χώρα. Επίσης θα πρέπει να αναφερθούμε στα προηγούμενα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Τουρκμενιστάν και να μην υποχωρήσουμε ως προσδοκίες που είχαμε από τη χώρα αυτή, γιατί είχαμε σημαντικά ορόσημα και γνώμονες που θα πρέπει να τηρήσει το Τουρκμενιστάν σε ό,τι αφορά την, α, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει να προβούμε σε μια αντικειμενική και αμερόληπτη αξιολόγηση τι χώρε αυτή ω προ τα ανθρώπινα δικαιώματα και φυσικά να δούμε πώ μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τι νέε δυνατότητε που μα δίνει η Συμφωνία εταιρική σχέση και συνεργασία. Και συμφωνώ με τον κύριο Πάσκου ότι θα πρέπει να περιλαμβάνουμε συμφωνία και μια ρήτρα που θα προβλέπει δυνατότητα αναστολή αυτή τη συμφωνία σε περίπτωση που δεν εφαρμόζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να εφοδιάσουμε τη συμφωνία με αποτελεσματικού μηχανισμού που μας, να μα εξασφαλίζουν την διαπίστωση πρόοδου και παρακολούθηση της πρόοδου του Τουρκμενιστάν ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όπως είπε και η συγκήτρια, οι συμβαστικές λύσεις που εκπονήθηκαν ε, πληρούν ε, τις προϋποθέσεις ε, και τις ανταπεξέρχονται προσδοκίες μας και την ευχαριστώ θερμά που έλαβε υπόψη και τις δικές μου τροπολογίες. Σας ευχαριστώ, κύριε Ολοκληρώνει τη συζήτηση η κυρία Γκόμες για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ήμουν μία από ε, όσους συνέταξαν περαιτέρω τροπολογίες και ευχαρίστω να δω τις, τροπολογίες, τις συμβιβαστικές που βρέθηκαν. Δεν μπόρεσα να τις δω και πραγματικά Είμαι μία από αυτού που συνέβαλαν περισσότερο με μετροπολογίε, αλλά που έχουν ε, σοβαρού δισταγμού για να συμφωνήσουν σε αυτή την έκθεση. Και γι' αυτό και θα ήθελα να ζητήσω από την εισηγήτρια και από τους Κιώδη να μου δείξουν τι ε, συμβιβαστικές και επίση και συμφωνώ με τα όσα είπαν διάφοροι συνάδελφοι, τι πληροφορίε που έδωσε η κυρία Κιλ Νίλσεν. Όντως υπήρξε αυτή η παρεμπόδιση ε, που δεν επέτρεψε σε διεθνεί ΜΚΟ να επισκεφθούν το Τουρκμενιστάν. Ευχαριστούμε κυρία Γκόμε. Ολοκληρώνεται τη συζήτηση τη Επιτροπή μα με την παρέμβαση τη κυρία Μικέζ από την Επιτροπή. Σας ευχαριστώ που μου επιτρέπετε να κάνω κάποια σχόλια. Εγώ δεν έχω δει ακόμα το κείμενο που προτείνεται με τις συμβιβαστικές και είναι λίγο δύσκολο να επεκταθώ, αλλά <coughs> θυμάμαι ότι προτείναμε τρία διαφορετικά είδη follow-up σε σχέση με τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπήρχε το θέμα διομετούς έκθεσης, ετήσιας συζήτησης και υπήρχε το θέμα του μηχανισμού παρακολούθησης. Από την άποψη της Κομισιόν δεν έχουμε κανένα πρόβλημα για ετήσια έκθεση. Ανέκαθεν το έχουμε επαναλάβει εδώ και στην Επιτροπή των Δικαιωμάτων και είμαστε έτοιμοι ετησίως να έρθουμε να σας ενημερώσουμε και να ε, σας ενημερώσουμε για τις ε, απόψεις μας για την ε, τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημοκρατία στο Τουρκμενικιστάν που ε, συμφωνώ απολύτω δεν είναι διόλου ικανοποιητική. Πόρο απέχει μάλιστα. Θα ήθελα λοιπόν να μπορέσω να δω το κείμενο γιατί είτε θα κάνουμε αυτό που ήδη λειτουργεί για την έκθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προετοιμάζουμε σε αιτήσια βάση και μπορούμε να φανταστούμε να έχουμε μια πιο λεπτομερή έκθεση για τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτή είναι η επιθυμία σας, δεν έχουμε πρόβλημα με αυτό. Διαφορετικά μιλάμε για ένα τελείως νέο μηχανισμό. Οπότε πιστεύω πως πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο και να δούμε ακριβώς τι σημαίνει κάτι τέτοιο. Ιδιαίτερα αν η κυρία Νικολάη θέλει να ευαθύνει, γιατί αν μιλάμε για ένα νέο μέσο, τότε έχουμε επιφύλαξη, διότι θα πρέπει να ελέγξουμε αν και κατά πόσο είμαστε μέσα στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεργασία του διοργανικού. Είμαστε στο πλαίσιο τη συνθήκη τη Λισαβόνα, αλλά η λήψη του κειμένου είναι δύσκολο να σα δώσω την οριστική μου γνώμη. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστούμε. Η εισηγήτρια, κυρία Νικολάη. Α, μια υπερώτηση. 30 δευτερόλεπτα η κυρία Χάουταλα. Ναι, συγγνώμη. Πρόεδρε, εγώ φαντάζομαι πως η Κομισιόν θα απαντήσει στην ερώτησή μου γιατί είναι πολύ σημαντική. Ήταν πολύ δύσκολο να έχουμε το κείμενο το οποίο συζητάμε και βρίσκουμε ότι έχει αποδυναμωθεί. Θέλω απάντηση. Θέλετε να συμπληρώσετε. Επιτροπή, μπορείτε να απαντήσετε στη συγκεκριμένη ερώτηση της κυρίας Χάουταλα. Ναι, καταρχήν το κείμενο που συζητάμε έχει ήδη ε, ε, υπογραφεί. Έγινε διαπραγμάτευση και έγινε ε, και υπογράφηκε. Δεν μπορεί να αναθεωρηθεί αυτό το κείμενο. Ε, υπήρχαν στοιχεία τα οποία συζητήθηκαν σε κάποια φάση και δεν τα βρίσκεται στο κείμενο. Τότε θα πρέπει να ανατρέξουμε στον άνθρωπο που ήταν επικεφαλή ε, των διαπραγματεύσεων πριν από 12 χρόνια. Μπορώ να το ελέγξω, αλλά το κείμενο είναι αυτό το οποίο διαπραγματευτήκαμε και υπογράψαμε τα κρατημέλη, το Κοινοβούλιο και το Τουρκμενιστάν. Ωραία. Η εισηγήτρια Νικολάη έχει το λόγο για να ολοκληρώσει. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταλαβαίνω πολύ καλά τις ανησυχίες των συναδέλφων, τις συμμερίζομαι. Ωστόσο, πιστεύω πως Είμαστε ενώπιον μιας πολιτικής εναλλακτική. Στην έκθεση έχουμε προβλέψει όλους τους μηχανισμούς επαλήθευσης, παρακολούθησης που μπορεί να χρησιμοποιήσει το Ευρωκοινοβούλιο. Ταυτόχρονα λυπάμαι γιατί βλέπω ότι οι τροπολογίες δεν διανεμήθηκαν στους συναδέλφους. Όμως, εάν δεν υπογραφεί αυτή η συμφωνία, θα συμβάλαμε στην τελμάτωση και στη διαιώνιση της κατάστασης στην περιοχή. Δεν θα μπορούσαμε δηλαδή να έχουμε διαφορετικά μια επικοδομητική προσέγγιση στην περιοχή αυτή. Φυσικά και μπορούμε να εφαρμόσουμε κυρώσεις, ε, να μιλήσουμε για τις δικές μας αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Ωστόσο, τέτοιες κυρώσεις μόνο να επιδεινώσουν την κατάσταση θα μπορούσαν, όχι να την βελτιώσουν. Στη συνέχεια, όσον αφορά την επιστολή των ΜΚΟ, ξέρω περί πρόκειται, ναι, πρόκειται για την είσοδο στο Καζακστάν και όχι στο Τουρκμενιστάν και το μόνο που γνωρίζουμε με τα βεβαιότητος εγώ προσωπικά είμαι νομικός, οπότε δεν εμπιστεύομαι τις μονομερείς δηλώσεις. Θα πρέπει πάντα να επαληθεύουμε τι συμβαίνει. Επαλήθευσα λοιπόν και αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι το Καζακστάν δεν εκχώρησε βίζα σε αυτές τις ΜΚΟ. Γιατί, υπό ποιες προποθέσεις, τι ακριβώς συνέβη, δεν μπορώ να ξέρω. Γιατί ε, και γι' αυτό το λόγο δεν θέλω να προβώ σε επικίνδυνες δηλώσεις. Δεν έχω αποδείξει τα χέρια μου για το τι ακριβώς, ακριβώς συνέβη. Και για την κυρία Χάουταλα να πω. Δυστυχώς όσοι σας εκπροσώπησαν στην τελευταία συνεδρίαση, οι σκιώδεις συζητητές ζήτησαν αυτή τη διατύπωση. Ίσως να μην τους εξηγήσετε ακριβώς τι θέλατε εσείς με αυτή την τροπολογία. γιατί δεν έγιναν τα πράγματα όπως τα θέλατε. Αλλά είμαι έτοιμη να το ξανασυζητήσουμε. Πιστεύω πως θα πρέπει να ευνοηθεί ένας επικοδομητικός διάλογος και όχι να μπλοκάρουμε τη συζήτηση. Τώρα, όσον αφορά την ίδια την έκθεση, να σας πω ότι ο μηχανισμός που προτείνεται με αυτή την έκθεση, που είναι ένας μηχανισμός τον οποίο επιτρέπει η συνθήκη της Λισαβόνας, το έχω παλιθέσει με την νομική υπηρεσία, αυτός ο μηχανισμός μας επιτρέπει να μεταβάλουμε την άκαμπτη θέση που είχαμε μέχρι τώρα και να είμαστε πιο δραστήριοι σε περιοχές όπου η συμβολή μας μπορεί να συμβάλλει στον εκδημοκρατισμό μια, έναν αγώνα που ταλανίζει αυτή τη χώρα, αλλά όχι μόνο αυτήν. Σας ευχαριστούμε κυρία Νικολάη. Όσον αφορά τις προθεσμίες, Η ψηφοφορία για την Επιτροπή προβλέπεται 25-26 Ιανουαρίου για να περάσει από την Σύνοδο του Μαρτίου, της 1ης Μαρτίου. Για το πολιτικό ψήφισμα δεν υπάρχει επιφύλαξη για το αν θα ψηφιστεί ακόμα και αν ε, εκφράστηκαν ανησυχίες, σχόλια κτλ. Όμως όσον αφορά την ψηφοφορία για την συμφωνία η εισηγήτρια επιμένει να γίνει και εμείς τη σεβόμαστε τη γνώμη τους. Α, όμως από όσα άκουσα δεν είμαστε βέβαιοι πως η πλειοψηφία των συναδέλφων ε, θα είναι υπέρ ε, τη υπερψήφισης της συμφωνίας. Τώρα, αν επιμείνει η, η, η εντάξει, εμεί θα το βάλουμε για ψηφοφορία, αλλά εγώ θα της πρότεινα να έρθει σε επαφή με τους Κιώδης για να βρεθεί κάποια συμβιβαστική λύση. Ή ίσως και να γίνει κάποια αλλαγή, ώστε να εγκριθεί το κείμενο, γιατί διαφορετικά Δεν είναι σκόπεμο, δεν ήθιστε να καταψηφίζετε μία τέτοιου είδους έκθεση. Ωραία λοιπόν, κλείνουμε τις εργασίες μας, θα τα ξαναπούμε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων μετά τα Χριστούγεννα στις 13 Ιανουαρίου, οπότε να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία, αν και ίσως τα ξαναπούμε κάτι δίαν πριν από τις γιορτές, αλλά όχι επισήμως. Ε, σας εύχομαι λοιπόν καλές γιορτές και θα τα πούμε τον επόμενο χρόνο στην Επιτροπή μας και στο Στρασβούργο για την Σύνοδο της Ολομέλειας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Λύεται τη συνεδρίαση.